η σημερινή συνεδρίαση είναι αφιερωμένη στη Σομαλία. Υπάρχουν πολλά από τα θέματα λοιπόν αυτά που μας αφορούν για την ε, ενέργεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της ε, πειρατείας και περιμένουμε συναδέλφους από την Επιτροπή Αλίας και την Επιτροπή Μεταφορών. Κύριο Σίμψον από την Επιτροπή Μεταφορών θα έλθει ε, μέσα σε λίγο χρόνο και η κυρία Φράγκα της από την Επιτροπή Αλίας σας πενθυμίζω ποιο είναι το... ποιες είναι οι τεχνικές ρυθμίσεις. Δεν θα έχουμε μετάφραση από τα μαλτέζικα, τα σλοβένικα, τα Λετώνικα, τα φιλανδικά και τα δανέζικα. Η συνεδρίαση μεταδίδεται στο διαδίκτυο όπως γνωρίζετε και όπως σας έλεγα προηγουμένως η μέση διάταξή μας αφορά απολύτως και αποκλειστικά την Σομαλία. Έχουμε δύο διαστάσεις, την καταπολέμηση της πειρατείας με την επιχείρηση Αταλάντη, Αταλάντα μάλλον, επικεφαλή στον άβαρχο, τον υπονάβαρχο Χάτσον που θα ακούσουμε σε λίγο και στη συνέχεια έχουμε τον Καρλ Χάτσεν, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος της ε, Σουηδίας, τον στρατηγό Ζωανά, ο οποίος είναι προσωπικός εκπρόσωπος του κυρίου Σολάνα για την Σομαλία και ο κύριος Ρότζερ Μουρ, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος της ε, ε Κομισιόν για το κέρας της Αφρικής. Αυτή τη στιγμή ξέρετε ότι εκτιλήσονται συζητήσεις για να δούμε ποια θα πρέπει να είναι συνέχεια που θα δώσουμε στις ε, συζητήσεις για την κατάρτιση ε, δυνάμεων ασφαλείας στην Σομαλία υπό την διοίκηση της μεταβατικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης στη Σομαλία. Αν δεν υπάρχουν λοιπόν ε, παρατηρήσεις μπορούμε να εγκρίνουμε την μέση διάταξη. Περνάω στο επόμενο θέμα, πρακτικά τη συνεδρία τη 30η Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου. Αν δεν υπάρξουν παρατηρήσει ω το τέλο τη συνεδρία, θα θεωρήσουμε ότι έχουν εγκριθεί τα πρακτικά αυτά. Και πρωτού δώσω το λόγο στον υπονάβαρχο Χάτσον. σα υπενθυμίζω ότι αύριο αποκινούμε την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Θα υποδεχτούμε στις 6.30 το απόγευμα τον Σουηδό Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Στόργολφς, ο οποίος θα μας παρουσιάσει τα αποτελέσματα του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών, που περιλαμβάνει και τους Υπουργού Άμυνας, που θα λάβει χώρα αύριο. Σας υπενθυμίζω ότι στις 30 Νοεμβρίου επίσης θα έχουμε και μία ε, ακρόαση που θα οργανώσουμε για το θέμα της μη διασποράς των ποινικών όπλων. Χωρίς να καθυστερήσω περαιτέρω, θα δώσω τον λόγο στον υπονάβαρχο Χάτσον, ο οποίος είναι επικεφαλής επιχειρήσεως Αταλάντα, που είναι μία, αν θέλετε, είναι η, μάλλον η πρώτη ναυτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας έξω από τις ακτές της ε, Σομαλίας. Ο Ναύαρχος Χάτσον εδώ και ένα χρόνο έχει φέρει σε πέρα σε ένα εξαιρετικό έργο. Είχα και εγώ ήδη την ευκαιρία πρόσφατα να βρεθώ στο Τζιμπουτί και να παρακολουθήσω τις ενέργειες αυτές. Προσκλήση του υπευθύνου των ναυτικών αυτών δυνάμεων και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον πώς, πόσο ικανοποιητικά γίνεται αυτή η επιχείρηση και πόσο υπερήφανα είναι τα πληρώματα για την ενέργεια αυτή η οποία είναι μια σαφής παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή αυτή. Σας δίνω τον λόγο λοιπόν. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, μέλη της Επιτροπής, καλησπέρα σας. Είναι τιμή και εμένα το ότι βρίσκομαι σήμερα εδώ πέρα και μπορώ να σας ενημερώσω για τα γεγονότα που αφορούν την επιχείρηση Αταλάντα που είναι η επιχείρηση καταπολέμησης πειρατείας στον κόλπο του Άντεν και στο δυτικό τμήμα του Ινδικού και τον Δεκέμβρη θα κλείσει ένα έτος. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου είχαμε 30 διαφορετικά πολεμικά πλοία τα οποία συμμετείχαν στις επιχειρήσεις και η διοίκηση ασκούνταν από το στρατηγείο στο Northwood και επιτόπου από ανωτά τους αξιωματικούς από την Ελλάδα, Ισπανία και την Ολλανδία. Το ΔΕΠ τελείωμα αποτελείται από αξιωματικούς από 16 χώρες, οπότε έχουμε μια πραγματικά ευρωπαϊκή γεύση στις ε, επιχειρήσεις. Να σας δώσω μια γενική εικόνα με βάση, ξεκινώντας βεβαίω από το γιατί ξεκίνησε αυτή η επιχείρηση. Θα θυμάστε πως ε, είχαν φτάσει το 2007 τα επίπεδα της πειρατείας σε απαράδεκτα επίπεδα και η διεθνής ε, κοινότητα και η ναυτική κοινότητα εξέφραζε όλο και πιο δυνατά τις ε, ανησυχίες τους καθώς δεν μπορούσαν να διέλθουν από αυτούς τους σημαντικότατους διάβλους. Το ΟΗΕ το 2008 αναγνώρισε την απειλή και πέρασε σύντομα σύντομα τέσσερα διαδοχικά ψηφίσματα που καλούσαν τη διεθνή κοινότητα να συντονίσει τις προσπάθειές της για να καταπολεμηθεί αυτή η δραστηριότητα. Αυξήθηκαν έτσι τα επίπεδα ανησυχίας και στο πρόγραμμα επισητισμού του ΟΗΕ που τότε έδινε σημαντική βοήθεια διατροφική Σομαλία υπό την προστασία διαφόρων διεθνών δυνάμεων. Η απειλή στα πλοία αυτά που επιχειρούν πολύ κοντά στι ακτέ ήταν πραγματική και μάλιστα ένα πρόγραμμα του προγράμματο αυτού, αν και φορτίου, ε, πειρατεία το 2007. Σωστά, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνώρισε τη σημασία αυτών των δύο στόχων, δηλαδή της καταπολέμησης πειρατείας, της προστασίας του υψηλιστικού προγράμματος και της προστασίας ευάλωτης ναυτιλίας προτάθηκε στα τέλη του περασμένου καλοκαιριού αυτή η ιδέα, επισήμως 20 Σεπτεμβρίου και η πρώτη επιχειρησιακή δυνατότητα επιτόπου είχε αναπτυχθεί στις 30 Δεκεμβρίου. Ε, πρόκειται για ένα επενεταίο επίτευγμα, καθώς ε, έγιναν όλα αυτά αποτελεσματικά, χωρίς πολύ πολύ φασαρία, με εύρωστη εντολή ξεκάθαρους κανόνες εμπλοκής και με επαρκές επίπεδο δυνάμεων. Η εξαίρετη δουλειά της Κομισιόν και των υπόλοιπων θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδήγησε σε μια νομική συμφωνία με την Κένια για να μπορέσουν να παραπενθούν στη Μομπάσα για δίκη οι συλληφθέντες, κάτι που αποτέλεσε ένα παράγοντα επιτυχίας της επιχείρησης και τώρα έχουμε μια επιχείρηση πλήρη και η δική μου η εντολή είναι σαφής. Είναι η ασφάλεια του προγράμματος του ε, ευσυτιστικού και των πλοίων που συνοδεύουν την ε, αφρικανική δύναμη στην Σομαλία. Επίσης την προστασία εμπορικών πλοίων ανεξαρτήτως ε, σημαίας και έχω στην διάθεσή μου δυνάμεις ευρωπαϊκής δυνάμεις για της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διαταράξω και όπου αυτό είναι δυνατόν να συλλάβω και τους πειρατές. Όπως ξέρετε επεκτάθηκε η εντολή μέχρι το τέλος του 2010 σε αρχές του έτους και δεν θα μου προξενήξει εντύπωση να επεκταθεί και παραπέρα. Ξεκινώντας με αυτές τις τρεις αποστολές λοιπόν, το ευσυντιστικό πρόγραμμα του ΟΗΕ ήταν πλήρως επιτυχημένη αυτή. Η πτυχή 50 πλοία συνοδεύτηκαν, πήγαν μένει οπομπή στην Σομαλία και δώσαμε 30.000 τόνους βοήθεια στο Μογκαντήσου και στις λοιπές πόλεις για παραπέρα διανομή 40 πλοία της Αφρικανικής δύναμης καλύφθηκαν για να δώσουν αυτή την υποστήριξη επιμελητία στην αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης και κανένα από τα πλοία αυτά υπό την προστασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν δέχτηκε επίθεση. Τα καθήκοντα αυτά, αν και αποτελούσαν υψηλή προτεραιότητά μας, ε, αποτελούν και σημαντικό φόρτο για τα στοιχεία που έχουμε στην διάθεσή μας και τα πλοία τα οποία μεταφέρουν αυτή την ε, βοήθεια είναι συχνά αργοκίνητα και διακινδυνεύουν έτσι και τα πολεμικά πλοία. Οι προσπάθειές μας ενισχύθηκαν με το να βάλουμε αγήματα επί των πλοίων αυτών, αλλά έπρεπε πρώτα απ' όλα να έχουμε διεθνή έγκριση και καθώς τα πλοία αυτά προέρχονται από κάποιες μικρές ε, χώρες, ε, Σιέρα Λεόν, ε, τις Κομόρες και μέχρι πρόσφατα ακόμα και τη Βόρεια Κορέα, Κορέα με συγχωρείτε, έκαναν δύσκολη αυτή την έγκριση, αλλά σημειώνεται πρόοδος και είμαι σίγουρος πως στο μέλλον θα έχουμε σημαντικές βελτιώσεις. Αυτή τη στιγμή απασχολείται ανά πάση στιγμή θα έλεγα μια μισή περίπου φρεγά για αυτό το καθήκον. Κατόπιν ανέφερα βεβαίως την προστασία της ε, ναυτιλίας. Πολλά πλοία πέφτουν θύματα πειρατείας και βεβαίως ε, η καταπολέμηση πειρατείας δεν ήταν τόσο εύκολη όσο θα θέλαμε. Εύκολο θα ήταν βεβαίως να σκεφτούμε πως ένα πλοίο το οποίο εφίσταται επίθεση με ρουκέτες και με άλλα μέσα θα μπορούσε να υποστεί μια ζημιά με, περιβαλλοντική, βεβαίως, με περιβαλλοντικό αντίκτυπο και πιθανή απειλή, ε, απώλεια ζωής. Συστάθηκε λοιπόν ένα κέντρο ασφάλειας της ναυτιλίας στον όρχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποστηρίζεται και από Ευρωπαίους αξιωματικούς του εμπορικού και του πολεμικού ναυτικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από άλλες χώρες σήμερα στο κοινό κέντρο επιχειρήσεων έχω εμπειρογνώμονε από την κοινότητα των δεξαμενοπλοίων, των κουρασγερόπλοίων, τη αναψυχή δηλαδή, και ακόμη και από την Ισπανική Ένωση Αλληλιαστών Τόνου. Όλοι αυτοί δίνουν συμβουλές στην ομάδα μου και, ακόμη σημαντικότερο, στα πλοία που πλέον στην περιοχή. Δίνουμε πολλές ε, συμβουλές. Μέτρα μη κινητικά αυτοπροστασίας, διαδικασίες ε, διέλευσης από τον κόλπο του Άντεν και επίκαιρες πληροφορίες. Τους ε, ενημερώνουμε για περιοχές οι οποίες έχουν εντοπιστεί υπό τα σκάφη. Οπότε υπάρχει ελεύθερη ροή πληροφοριών. Το κέντρο βεβαίως είναι στο διαδίκτυο με πρωτόκολλα ασφαλείας ανάλογα με αυτά του e-banking και επιτρέπεται έτσι να χρησιμοποιηθεί και από αυτούς που δρούν επιτόπου στον κόλπο του Άντων. Τα πλοία τα οποία, του Άντεν, τα οποία είναι αργοκίνητα και έχουν χαμηλά το κατάστρωμα, μεταφέρουν φορτίο υψηλής ε, αξίας, θεωρούνται πλοία υψηλού κινδύνου και όπου μπορούμε τα συνοδεύουμε από τις περιοχές μεγάλης απειλής. Και αυτές ε, τις πληροφορίες τις δίνουμε και στο ΝΑΤΟ που έχει παρουσία επιτόπου για να ξέρουν όλοι που είναι αυτά τα πλοία υψηλού κινδύνου και να μπορούμε όλοι να έχουμε το νου μας. Όσον αφορά τον συντονισμό τώρα μεταξύ του στρατιωτικού και του πολιτικού σκέλους. Νομίζω ότι έχουμε ένα παράδειγμα βέλτιστων πρακτικών και οι διαδικασίες μας εγκρίθηκαν πρόσφατα από τον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας ως ε, το βασικό μέσο συνεννόηση των πλοίων στην περιοχή. Λίγα από τα πλοία τα οποία ακολούθησαν τις συμβουλές μας τα κατέλαβαν πειρατές και τα πλοία τα οποία θεωρήσαμε ευάλωτα τα συνοδεύσαμε από το διάβλο και πάλι κανένα από αυτά δεν κατελήφθη τους πειρατές. Οπότε λειτουργεί το σύστημα αλλά σημαίνει πως θα πρέπει να μας ειδοποιούν τα πλοία και παρά την τεράστια δημοσιότητα του ζητήματος της και τις τραυματικές συνέπειες μιας πειρατείας Ακόμα έχουμε πολλά πλοία που επιλέγουν να μην έρθουν σε επαφή μαζί μας και προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε. Τα κράτη-μέλη πρέπει να επαναλάβουν στις εθνικές ναυτιλιακές οργανώσεις την σημασία του κέντρου μας και να ενθαρρύνουν το να μας ειδοποιούν τα πλοία όταν περνάνε από τον Ινδικό. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε όλες τις επιθέσεις στα πλοία, αλλά μπορούμε οπωσδήποτε να βοηθήσουμε τα πλοία να μειώσουν την πιθανότητα επιτυχίας των επιθέσεων. Όπως σας είπα, στόχος μου είναι να αποτρέψουμε να διαταράξουμε τις επιθέσεις και να συλλάβουμε τους πειρατές όπου αυτό είναι δυνατόν. Και πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός για να βρεθούν οι ύποπτοι ενώπιον ενός δικαστηρίου. Η βασική ευθύνη για αυτό στο διεθνές δίκαιο βεβαίως βρίσκεται, την επομίζεται η χώρα η οποία κάνει την σύλληψη και θα πρέπει τα κράτη-μέλη να δουν, ε, μεμονωμένα να δουν εάν διατεθειμένα να φέρουν αυτούς τους ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να δικαστούν. Κατά κανόνα δεν το κάνουν αυτό, οπότε έχουμε μια συμφωνία με την Κένια για μεταφορά των υπόπτων εκεί πέρα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Ο σύνδεσμος με την πολιτική πτυχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάρα πολύ μεγάλος και είμαι τυχερός... Ε, από την ομάδα στην Γενική Διεύθυνση 8, τι εξωτερικέ σχέσει και την υπόλοιπη Κομισιόν αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι του αποτρεπτικού μας ρόλου. Βεβαίως, οι επιχειρήσει γίνονται μόνο με σκάφη και αεροσκάφη, δεν μπορεί να γίνει από τον Όρκο. οπότε ανά πάση στιγμή πρέπει να βρίσκονται τέσσερα πλοία εμπλό και τρία αεροσκάφη αεροναυτική συνεργασία για την περιπολία. επίση για να υπάρξει συντήρηση, αλλαγή των πληρωμάτων και ανεφοδιασμός ε, σημαίνει πω θα έχουμε ανα πάσα στιγμή στο θέατρο των επιχειρήσεων 5 ή 6 πολεμικά πλοία. Και τα έχουμε αυτά. Τα κράτη-μέλη μα έδωσαν πάρα πολλέ μονάδε και καθ' όλη τη διάρκεια του 2009 είχαμε τι απαραίτητε δυνάμει. Ενισχύουμε τώρα τι δυνάμει μα για το 2010 και είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξο για το ότι θα έχουμε επαρκή αριθμό πλοίων και αεροσκαφών για το επόμενο έτος. Ας δούμε τώρα σύντομα τους δύο βασικούς ε, τομεί οποίους επιχειρούν οι πειρατές. Πρώτα απ' όλα ο κόλπος του Άντεν. Είχαμε σειρά επιθέσεων, σοβαρών επιθέσεων το 2008 και το πρώτο εξάμεινο του 2009. Τουλάχιστον 12 πλοία κατελήφθησαν και 42 άγριες επιθέσεις ε, συνέβησαν. Του τελευταίου μήνε είχαμε σημαντική πτώση τη δραστηριότητα με ελάχιστε επιθέσει και κανένα πλοίο δεν έπεσε στα χέρια των πυρετών από τα μέσα του Ιουλίου. Γιατί αυτό. εμεί θεωρούμε πω υπάρχουν τρει λόγοι. Πρώτα απ' όλα το επίπεδο συντονισμού, η στρατιωτική παρουσία και η γενικότερη παρουσία των πλοίων μα είναι πολύ υψηλότερη από ότι ήταν πριν το 2008 και 2009. Έχουμε καλό συντονισμό και ακολουθούν μέτρα αυτοπροστασία στα εμπορικά πλοία. Ο συντονισμός τους επιτρέπει να έχουν πληροφορίες εγκαίρως όταν βλέπουμε ύποπτη δραστηριότητα. Οπότε έχουμε αποτροπή. Ο καιρός στον κόλπο του Άντεν αυτή τη στιγμή ευνοεί άλλες εγκληματικές δραστηριότητες. Π.χ. λαθρεμπόριο ανθρώπων από την Σομαλία προς την Ιεμένη που έχει αυξηθεί πολύ τους τελευταίους μήνες. Για τους εγκληματίες που κάνουν αυτές τις ε, επιχειρήσεις, η δυνατότητα να μεταφέρουν ανθρώπους έχει μικρότερο κίνδυνο και υψηλότερη ανταμοιβή, οπότε πέρασαν σε αυτή τη δραστηριότητα. Και βλέπουμε βεβαίως περιοχή του Πούντ ε, οι αρχές από ξηράς ε, έχουν αυξήσει την παρουσία τους, οπότε μειώνονται έτσι οι επιθέσεις. Δεν υπάρχει όμως περιθώριο για χαλάρωση. Επαναλαμβάνω πως μιλάμε για παγκόσμια αρτηρία της ναυτιλίας δεν πρέπει να ε, ε, αναζωπηρωθεί το φαινόμενο και πρέπει να αντιδράσουμε άμεσα. Πρέπει να εξορροπήσουμε επίσης ε, τις δυνάμεις μας στον κόλπο του Άντεν και στην Σομαλία. Για την Σομαλία τώρα τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων ήταν πιο δραματικά. 8 πλοία κατελήφθησαν. Είχαμε 21 βεβαιωμένες επιθέσεις, 21. Όπως σας είπα, οι επιτυχίε μας στον κόλπο του Άντεν έκαναν τους πειρατέ να επανεξετάσουν την τακτική τους και μετακινήθηκαν νότια στον Ινδικό ωκεανό. Έφτασαν μέχρι και τις Αιχέλε και ακόμη πιο νότια τις τελευταίε εβδομάδες και έχουν κάποια πλοία που τους τροφοδοτούν είτε είναι πλοία τα οποία έχουν καταλάβει και είναι λάτζες, είτε κάποια αλλιευτικά σκάφη, καθώς αφενός κάνουν ελαφραλία και την επόμενη μέρα κάνουν πειρατεία, για να μπορέσουν να φτάσουν στους διάβλους της ναυτιλίας. Πρόκειται για άτομα απελπισμένα και δεν έχουν πρόβλημα να μένουν σε ένα σκάφος ανοιχτό επί στον ωκεανό. Και βέβαια η ζωή τους έχει μικρή αξία, ειδικά για τα αφεντικά τους στην ξηρά. Κάποια στιγμή είχαν φτάσει 18 πλοία να είναι εγκυροβολημένα και περίμεναν την λήξη των διαπραγματεύσεων για τα λίτρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 10 πλοία στα χέρια των πειρατών με 244 άτομα μέλη του πληρώματος στα χέρια τους. Να σας υπενθυμίσω όμως το μέγεθος του ωκεανού. Έχουμε 1,5 εκατομμύριο τετραγωνικά χιλιόμετρα Δύο τρίτα δηλαδή το μέγεθος των ΙΠΑ, το δε με... μέγεθος της ακτογραμμής στα ανατολικά της ε, Σομαλίας είναι 2.800 χιλιόμετρα. Δηλαδή από τις Βρυξέλλες θα φτάναμε στην Μόσχα. Οπότε ένα αεροσκάφος που εντοπίζει μια βάρκα και επιρεχειρούν από το Τζιμπουτί, τη Μομπάσα και τις Ειχέλες τα αεροσκάφη μας. Ένα σκάφος λοιπόν που εντοπίζει μια βαρκά μεγαλύτερο σκάφο των πειρατών αναμένει μία και δύο ημέρε για να το πλησιάσει ένα πολεμικό πλοίο και βέβαια μέχρι τότε έχουν φύγει οι πειρατέ. Οπότε θα αναφέρω τρία πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μόνιμη παρουσία στην λεκάνη της Ομαλίας από τα μέση Αυγούστου. Βεβαίως ο Μουσώνας παραμένει προβλέψιμος και σταματάει στα μέση Σεπτεμβρίου, οπότε εμείς έχουμε τοποθετήσει μονάδες μας όσο δυνατόν καλύτερα. Έχουμε συνεργαστεί με το Λουξεμβούργο που έχει μισθώσει πολιτικά σκάφη ναυτικής επιτήρησης ε, τα οποία τοποθετήσαμε στις Σεϊχέλες οπότε καλύψαμε το νοτιοανατολικό τεταρτημόριο της λεκάνης της, των Σεϊχελών αποτελεί πολύ σημαντικό στοιχείο και μας έχει δώσει μεγάλες δυνατότητες. Δοκιμάσαμε να τοποθετήσουμε πλοία από εκεί που ξέρουμε ότι επιχειρούν οι πειρατές και κοντά σε Σεϊχέλες. Τα στρατόπεδα όμω των πειρατών μετακινούνται, γνωρίζουμε τουλάχιστον 70 από αυτά, καταλαμβάνουν πλοία και αλλιευτικά σκάφη, σα το είπα, οπότε είναι αδύνατον να κλείσουμε όλη αυτή την ακτογραμμή για να έχουμε κάποιο επίπεδο επιτυχία, αλλά προσπαθούμε. Μόλον τούτο, δεν πρέπει να δούμε μονάχα την αρνητική πλευρά, την απώλεια αυτών των πλοίων που δείχνει ότι δεν έχουμε επιτύχει το στόχο μας. Έχουμε συλλάβει 36 πλοία πειρατών στις ακτές της Σομαλίας. Πολλά από αυτά έχουν βυθιστεί και οι πειρατές έχουν συλληφθεί, μεταφερθεί στη Σομαλία και μετά στην Κένια για δικαστικές ενέργειες. 14 άμεσες επιθέσεις έχουν αποκρουστεί από τις δυνάμεις μας, έμεσα ή άμεσα, αλλά έχουν αλλάξει και οι τακτικές που ακολουθούν οι πειρατές. Όπως ξέρετε, έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο εξελιγμένη δράσης για να αντιμετωπίζουν μεγάλα πλοία πετρελοφόρα που δεν έχουμε δει στο παρελθόν. Το πιο σημαντικό στοιχείο βέβαια είναι ότι τα πλοία τα οποία καταλαμβάνονται στις ακτές της Σομαλίας δεν άκουγαν τις συμβουλές μας που ήταν και πάρα πολύ σαφείς για τα πλοία που πλέουν γύρω από το κέρα της Αφρικής. Επομένως, αυτά τα πλοία φταίνε σε κάποιο βαθμό για το γεγονός ότι συλλαμβάνονται. Οι πειρατέ έχουν αυξήσει την περιοχή δράση του και δύο πλοία έχουν τώρα καταληφθεί εκτό από την περιοχή δράση τη Αταλάντα. Είναι απαραίτητο λοιπόν να ακούν τι συμβουλέ μα τα πλοία και να μην προσπαθούν να λοξοδρομήσουν ή να βρουν πιο σύντομε διαδρομέ, γιατί αυτό σημαίνει ότι είναι υπεύθυνοι για την τύχη του μετά. Θέλω να τονίσω επίση ότι έχουμε πολύ καλέ σχέσει με τι αρχέ τη περιοχή του Πούντ και του Σάσο και με τι αρχέ στην Μπερμπέρα τα γαλλικά, ισπανικά και γερμανικά πλοία έχουν όλα συμμετάσχει σε κοινέ ενέργειε στι περιοχέ αυτέ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε λοιπόν με αποφασιστικότητα τι ενέργειέ μα, γιατί με τον τρόπο αυτό μπορούν οι ναυτικέ δυνάμει να μπορέσουν να εξασφαλίσουν ότι θα υπάρξει και μια πιο μόνιμη οικοδόμηση τάξη και νόμου στο μέλλον. Ο διάλογος αυτός λοιπόν είναι θεμελιώδης για να επιτύχουμε αυτό το στόχο. Δεν είμαστε μόνοι όμως. Δεν, είμα... δεν δρούμε μεμονωμένα για να αντιμετωπίσουμε την πειρατεία. Έχουμε ναυτικές δυνάμεις από 20 χώρες, οι οποίες κατά καιρό έχουν συμμετάσχει. Η Ινδία, Κίνα, Μαλαισία, Ιαπωνία, Ρωσία είναι ενεργέ αυτή τη στιγμή. Ο συντονισμό λοιπόν όλων αυτών των ναυτικών δραστηριοτήτων είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι ένα τομέα όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παίξει ένα προεξάρχοντα ρόλο, ιδίω στην περιοχή αυτή. Έχουμε κάνει συναντήσεις, έχουμε ανταλλάξει τα διδάγματα τα οποία έχουμε συλλέξει και υπάρχει τώρα καλύτερη επαφή μεταξύ όλων των πλευρών. Μετά από μια επίσκεψη στο Πεκίνο έχουμε συμφωνήσει με την Κίνα για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ε, συνεργασία μας μεταξύ κινέζικων και ευρωπαϊκών δυνάμεων στον κόλπο του Άδεν. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Επομένως βελτιώνουμε τις ικανότητές μας επιχείρηση είναι ήδη πάρα πολύ αξιόλογη, γιατί έχουμε αντιμετωπίσει πάρα πολύ σημαντικές στρατηγικές ευκαιρίες τα τελευταία, τους τελευταίους μήνες. Το ΝΑΤΟ <clears throat> έχει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Από τις 17 Αυγούστου ξεκίνησε η δράση η κοινή με το ΝΑΤΟ. Μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ προσπαθούμε να είμαστε συμπληρωματικοί. Ο στόχος μας δεν είναι να ανταγωνιστούμε οι μεν τους δε, Μέχρι στιγμή ήταν πάρα πολύ αποτελεσματική αυτή η συνεργασία. Μπορούμε από κοινού να βρούμε τρόπου να χρησιμοποιήσουμε τι ιδιαίτερε δεξιότητε που μπορεί να έχει ο κάθε φορέα για την επίτευξη του κοινού στόχου και προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι μιλάμε με την ίδια <clears throat> γλώσσα. Ιδίω όταν επικοινωνούμε με τι αρχέ τη Ομαλία. Η συλλογή πληροφοριών επίση είναι πάρα πολύ σημαντική και κάνουμε ό,τι μπορούμε να μπορούμε να καταλήγουμε σε κοινή εικόνα για τι επικίνδυνε και ύποπτε δραστηριότητε σε όλη αυτή την περιοχή. Τα ε, αεροπλάνα περιπολίας που πετούν με τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΝΑΤΟ δίνουν στοιχεία για όλους τους στην περιοχή της ε, Σομαλίας. Μαζί λοιπόν με την ε, Αμερικανική δύναμη η οποία προέρχεται από το υπάρχει μια στενή συνεργασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσπαθήσει να αναπτύξει συστήματα επικοινωνία για όλου του χρήστε, ένα ασφαλέ σύστημα που λέγεται Mercury, το οποίο επιτρέπει τα δεδομένα αυτά να ανταλλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια. Ιδίω η πρώτη ανείχνευση επικινδύνων ή ε, υπόπτων πλοίων. Δεν έχει νόημα να λέει ένα ιαπωνικό αεροπλάνο ότι υπάρχει κάτι μάλλον πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα και ένα Ιαπωνικό αεροπλάνο να δίνει σαφείς πληροφορίες σε ευρωπαϊκές αρχές, σε αρχές του ΝΑΤΟ για τα θέματα αυτά. Ξέρουμε ότι το θέμα της πειρατείας δεν θα λυθεί με το να τρέχουμε σαν τρελή στην περιοχή της Σομαλίας και στον κόλπο του Άδεν χρειάζεται μια πιο μόνιμη αντιμετώπιση. Η δική μου επιχείρηση είναι απλώ ε, μια συνιστόσα μια επιχείρηση, που είναι κυρίω μια επιχείρηση στην ξηρά. Εργαζόμαστε με φορεί κατά τη πειρατεία όπω είναι ο Διεθνή Οργανισμό και φορεί τη Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν συγκληθεί για να αντιμετωπίσουν το δυναμικό να υπάρχει καλύτερη αντιμετώπιση σε στρατηγικό τομέα και προσβλέπω σε περαιτέρω συζητήσει σε σχέση με τα θέματα αυτά στη συνέχεια του απογεύματο. Έχουμε Πάντως, ε, διαπιστώσει ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε και αναθεωρείται η εντολή μας για να περιλάβει και αυτές τις νέες στοιχείες. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε όμως τις προσδοκίες. <clears throat> Μέσα στις δομές που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μεγάλο περιθώριο ελιγμού. Υπάρχει έλλειψη υποδομών ε, στις ακτές για να εκμεταλλευτεί τι δυνατότητε που αναπτύσσουμε, δεν θα πρέπει να δρούμε μονάχα σε ένα συμβολικό επίπεδο, θα πρέπει να δράσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να δώσουμε πραγματικό άμεσο αποτέλεσμα. Τέλος, θέλω να σας πω ότι παρά όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει στις τελευταίες εβδομάδες, η ευρωπαϊκή επιχείρηση Αταλάντα λειτουργεί πολύ καλά. Είναι σαφή η εντολή τη και την εκπληρώνουμε. Έχουμε καλό προσωπικό, έχουμε καλή διοίκηση, έχουμε αποτελεσματική και παραγωγική σχέση με όλους τους εταίρους μας Και είμαστε έτοιμοι για νέες προκλήσεις και αλλαγές. Θα υπάρξουν τέτοιε αλλαγές γιατί τα γεγονότα μπορεί να στραφούν εναντίον μα, στις ακτές της Σομαλίας. Αλλά πιστεύουμε ότι με τις δυνατότητες που έχουμε μπορούμε πράγματι να εκπροσωπήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση με έναν τρόπο που θα είναι αποτελεσματικός και υπερήφανος. Αυτά λοιπόν και είμαι έτοιμος να απαντήσω οποιοδήποτε ερώτημα. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτή. Ήταν πάρα πολύ πλήρης και πραγματικά πάρα πολύ πολύτιμη. Ε, επί του συνόλου ε, της ε, επιχείρησής σας. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον πρόεδρο Σίμψον ε, και στον αντιπρόεδρο. Αλλά θα ήθελα να πω το εξής. Όσον αφορά το θέμα της πειρατείας, Πώς βλέπετε ότι, υπάρχει, ότι συνδέεται αυτό με την πολιτική αστάθεια στη Σομαλία, δεδομένου ότι οι βάσεις της πειρατείας ε, κυρίως ε, στο Πούντ ε, από εκεί προέρχονται και υπάρχει βέβαια και το πρόβλημα των Ισλαμιστών που δραστηριοποιούνται και σε άλλες περιοχές της Σομαλίας. Μήπως υπάρχουν κάποιες συνδέσεις μεταξύ αυτών των δύο φαινομένων. Και επίσης, επειδή προσφάτως ήμασταν εκεί, Υπήρχαν κάποιοι πειρατέ, οι οποίοι αντί να κάνουν πειρατεία εναντίον ε, των εμπορικών πλοίων, φορτηγών πλοίων ή άλλων, ε, ουσιαστικά διαφοροποιούν τις δραστηριότητές τους ε, στο εμπόριο ανθρώπων, στον κόλπο του Άντεν. Οπότε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα φαινόμενα έχετε, την, ε, έχετε σκεφτεί πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό και αν ναι πώς. Αυτά τα δύο λοιπόν ήθελα να πω, αλλά θα ήθελα να δώσω πρώτα το λόγο στον πρόεδρο Σίμψον, που, τον πρόεδρο της Επιτροπής ε, Μεταφορών και Τουρισμού, ε, με την οποία συνδιοργανώνουμε την σημερινή ακρόαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη που άργησα λιγάκι και έχασα την αρχή της παρουσίασης του υποναβάρχου Χάτσον. Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία τα οποία ε, μου έκαναν εντύπωση σε σχέση με αυτά που είπατε. Καταρχάς ε, θα ήθελα να πω, επειδή είμαι από την ε, βορειοδυτική ε, Αγγλία και επειδή έχουμε πάρα πολύ σημαντικές ναυτικές παραδόσεις εκεί, ε, θα, καταγνωρί... θα γνωρίζετε βεβαίως ότι έχουμε ιδιαίτερη ανησυχία για το ζήτημα της πειρατείας ε, που έχει ε, επικεντρωθεί πλέον στο κέρας της Αφρικής. Ακούγοντάς σας αναρωτιέμαι εμείς στην Επιτροπή Μεταφορών που συνεργαζόμαστε με τους συναδέλφους μας ε, στην Επιτροπή αυτή, πώς μπορούμε να συνεργαστούμε. Αν κατάλαβα καλά είπατε ότι μερικά ε, εμπορικά πλοία ουσιαστικά αγνοούν την καθοδήγησή σας και ουσιαστικά διακινδυνεύουν την κατάστασή τους. Αυτό μου φαίνεται πραγματικά απίστευτο. καταλαβαίνω βέβαια ότι μάλλον θα συμβαίνει και δεν ξέρω βέβαια τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ε, για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε σε πλαίσιο, στο πλαίσιο της ε, Διεθνούς Οργάνωσης Ναυτιλίας, ε, να προσπαθήσουμε να ενθαρρύνουμε τους πλειοκτήτες, να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση και να ακολουθήσουν τις συμβουλές σας δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο περίεργο να μην ακολουθούν ε, τις συμβουλές μας ε, τα πλοία σε τόσο επικίνδυνα ύδατα. Κάτι ακόμη αφορά το θέμα των ε, κυρίων πλοίων της περιοχής. Είπατε σε κάποια στιγμή της παρουσίασής σας ότι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε ήταν η έλλειψη της ε, ύπαρξης των ε, των πλοίων αυτών. Δηλαδή είπατε ότι υπήρχε, ότι υπήρχε αυτό το πρόβλημα και θα ήθελα να μου το εξηγήσετε. Υπήρχε επίσης το θέμα των ιδιωτικών ε, σκαφών που επίσης είναι αντικείμενο ε, πειρατείας προφανώς. Οπότε αναρωτιέμαι πώς μπορούμε να ε, τους βοηθήσουμε, δηλαδή τα ιδιωτικά σκάφη, τα σκάφη αναψυχής, να ε, μην πηγαίνουν σε αυτή την περιοχή, ώστε να μην είναι στόχοι της πειρατείας, γιατί ε, καταλαβαίνω ότι Και επειδή ήμουν στι ειδικέ δυνάμει, θα ήθελα να πω και το εξή. Ειδικότερα για, τις, τα ιδιωτικά σκάφη, ειδικότερα για την πειρατεία εναντί αυτών των σκαφών, το δίλημα που υπάρχει είναι το εξή. Είτε πηγαίνει κανείς ε, και συμμετέχει με αποτέλεσμα να πληγεί, είτε ε, καταλήγουν ε, σε ομοιρία. Οπότε πρέπει να δούμε, χωρίς να μπούμε εντάξει, σε πάρα πολλέ λεπτομέρειε, είναι να δούμε πώ θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα με τι ειδικέ δυνάμει, ε, με τι δυνάμει ε, που θα μπουν στο σκάφος για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Οπότε, θα ήθελα να πω στον υπονάβαρχο ότι θα του ήμουν ιδιαίτερος ευγνώμων αν μπορούσε και ελπίζω και οι υπόλοιποι συνάδελφοι να συμφωνήσουν, ε, να διαβιβάσει τις ευχαριστίες Επιτροπής Μεταφορών ε, σε όλους όσους, ε, σε όλη σας την ομάδα που κάνουν μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά, υπό πολύ δύσκολες συνθήκες, για να μπορεί να είναι ασφαλή η ναυτιλία στην περιοχή. Θα ήθελα λοιπόν να διαβιβάσετε τις ευχαριστίες αυτές και θα σας ήμουν ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε Σίμψον. Και βεβαίω και τι δικέ μα ευχαριστίε θα θέλαμε να μεταβιβάσετε. Ο Αλέν Καντέκ ε, για την ε, Επιτροπή Αλία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν σας ευχαριστώ να μου που δεχτήκατε αυτή την πρόσκληση. Και χαίρομαι που έγινε αυτή η κοινή συνεδρίαση με την Υποεπιτροπή Άμυνας αλληλείας και μεταφορών. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να έχουμε μια κοινή αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Είναι η καλύτερη λύση λοιπόν. Θα ήθελα καταρχήν να ζητήσω συγγνώμη εξ ονόματος της κυρίας Κάρμεν Φράγα, η οποία δεν μπόρεσε να είναι παρούσα σήμερα, γιατί είναι στο αεροπλάνο που τη μεταφέρει στο Ριτσίφ για να συζητήσει τις αλληλευτικές συμφωνίες για τον γαλαζόπτερων τόνων. Θα θυμόσαστε, πρόεδρε Ντάουνσον και πρόεδρε Σίμψον, ότι τονίσατε την ανάγκη να υπάρχει αυτή η μονάδα, η ναυτική δύναμη στην Αταλάντα, της Αταλάντα. Προφανώς ο τομέας αλίας σας ευχαριστεί που υπάρχει αυτή η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην, στον χώρο αυτό. Θα πρέπει να σκεφτούμε λιγάκι καλύτερα πώς θα λειτουργήσει η Αταλάντα. Μιλάω για τα ψάρια τώρα, δεν μιλάω για, για πειρατεία μόναχα. Πώς θα λειτουργήσει λοιπόν η Αταλάντα σε σχέση με την ιδέα ότι της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιήσει περισσότερο ε, πολεμικά πλοία της ε, Γαλλίας, ενώ η ισπανική ε, άποψη είναι να δοθούν σε ιδιωτικές εταιρείες τα θέματα άμυνα στην περιοχή. Έχουμε μια σαρανταριά περίπου πλοίων που αλλιεύουν τόνο, που βέβαια είναι κυρίως ισπανικά και γαλλικά, μερικά ιταλικά κτλ, αλλά κυρίως γαλλο-ισπανικά. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον για τον αλληλευτικό στόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι κάτι λοιπόν το οποίο είναι σαφές, ότι τα αλληλευτικά μας πλοία είναι ευάλωτα. Καταρχήν, είναι εύκολο να ανέβει κανείς σε αυτά τα πλοία, έχουν χαμηλά καταστρώματα και επίσης στη διάρκεια της διαδικασίας αλλίας είναι ακίνητα τα πλοία αυτά. Εκεί λοιπόν που αλλιεύουν τον τόρο μπορεί να τους αλλιεύσουν πειρατές. Επίσης, 75% της περιοχής της ε, αλίας που ασκούν αυτά τα πλοία είναι μέσα στην ε, περιοχή που καλύπτει η επιχείρηση Αταλάντα, δηλαδή της περιοχής κινδύνου. Οι πειρατές, όπως είπατε και εσείς, φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή έχουν κατέβει πιο πολύ προς τα νότια, προς τις Σεϊχέλες, για να πιάσουν τα πλοία τα οποία πηγαίνουν στις Σεϊχέλες και αυτό ίσως απαιτεί μια νέα ανάπτυξη των δυνάμεων. Σήμερα λοιπόν <clears throat> οι δυνάμεις της Αταλάντα εξασφαλίζουν σε μεγάλο βαθμό την προστασία αυτών των πλοίων, αλλά δεν δίνουν μια βέλτιστη προστασία των αλλιευτικών πλοίων, που πράγματι ως εκ της φύσης τους είναι πάρα πολύ ευάλωτα. Η προστασία τώρα των αλλιευτικών πλοίων με δυνάμεις που είναι πάνω σε αυτά τα πλοία και με οπλικά συστήματα, ίσως είναι η μόνη λύση και αυτή πιστεύω ότι είναι πράγματι συμβατή με την επιχείρηση Αταλάντα. Υπάρχει λοιπόν μια συμπληρωματικότητα μεταξύ των δράσεων αυτών και της Αταλάντα. Πρέπει καταρχήν να υπάρχει μια ταχεία διάδοση των δεδομένων για την παρουσία πειρατών και επίσης σημαντική είναι και η συμβολή των εναρίων δυνάμεων για να μπορέσει να υπάρξει αυτή, αυτός ο εντοπισμός των πειρατών και επίσης η δράση των διοκτικών και αστυνομικών δυνάμεων μετά τον εντοπισμό των πειρατών. Όλα αυτά λοιπόν μπορούν να βοηθήσουν να υπάρχει καλύτερη αποτελεσματικότητα της Αταλάντα σε ό,τι αφορά τα αλληλευτικά σκάφη και πιστεύω ότι θα είναι σημαντικό η εντολή της Αταλάντα να αναφέρεται σε τρία σε τρεις κατηγορίες. <clears throat> τα πλοία τα οποία είναι ευάλωτα κατά τη διάρκεια τη διέλευσής τους προς τον, από τον ε, κόλπο του Άντεν, αυτά τα οποία είναι επίσης ευάλωτα στην έξοδο τους από τον ε, κόλπο αυτό και φυσικά και τα αλλιευτικά πλοία και κυρίως τα πλοία τα αλληλευτικά επειδή είναι πάντα σε αυτή την περιοχή και είναι αργοκίνητα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντιμετωπιστούν σε χωριστή κατηγορία. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρχει ένα χωριστό πρωτόκολλο, καταρχήν να υπάρχει μια ομάδα προστασία στα πλοία αυτά πάνω στα πλοία όπως είπα, δεύτερον να ενσωματώνται καλύτερα σε δράσεις όπως η επιχείρηση τα Αταλάντη και να υπάρχει μια ειδική κρυσάρα σε σχέση με το πόσο ευάλωτα είναι όλα αυτά τα πλοία που να εφαρμόζεται ιδιαίτερα στα πλοία τα αλληλευτικά και επίσης να υπάρχει μια καλύτερη παρακολούθηση των πλοίων τα οποία είναι ύποπτα για άσκηση πειρατείας, γιατί αν περιμένουμε απλώς μια επιβεβαίωση αυτό μπορεί να πάρει πάρα πολύ χρόνο. Καλύτερη πληροφορία για, στα πλοία τα αλληλευτικά για τους διαδρόμους των περιπολιών και τέλος η επιτάχυνση της ε, έγκρισης της σύμβασης του Montego Bay σε σχέση με τις ενέργειες κατά της πειρατείας και της ε, Αταλάντα συγκεκριμένα. Αυτά ήθελα να σας πω λοιπόν. Και ένα τελευταίο ερώτημα θέλω να σας θέσω. Από ό,τι κατανοήσατε, είναι μια δραστηριότητα που ενδιαφέρει πάρα πολύ την Ευρώπη, ιδίω στην περιοχή αυτή. Θα ήταν ίσως χρήσιμο να υπάρξει και μια συμμετοχή στρατιωτικών δυνάμεων, ναυτικών δυνάμεων από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επιχείρηση Αταλάντα για να εξευρωπαϊστεί ακόμα περισσότερο αυτή η διαδικασία. Αυτό ήταν λοιπόν το ερώτημα που ήθελα να σας θέσω. Euh, Ευχαριστώ. Τρει συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Θα του δώσω το λόγο πρώτα και μετά θα απαντήσετε σε όλε τι ερωτήσει. Ο κύριο Καλέρα από το ΕΛΚ. Äh, ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και κύριε Νάβαρχε για τις αναλυτικές σας εξηγήσεις. Πρώτα απ' όλα μια σύντομη ερώτηση για το θέμα Ευρωπαϊκή Ένωση ΝΑΤΟ. Είπατε πως είναι εξαίρετη η συνεργασία. Πολιτικά θα έλεγα πως δόξα το Θεό λειτουργεί, αλλά ακόμη καλύτερο θα ήταν να έχουμε μόνο έναν από τους δύο οργανισμούς ε, ε, οργάνωση, να ασχολείται με την οργάνωση και τον συντονισμό εκεί πέρα. Για να μην ε, κάνουμε το ίδιο πράγμα από δύο πλευρές. Ένα ερώτημα. Με ποια κριτήρια μετράτε την επιτυχία της αποστολής. Είναι επιτυχία η συνεργασία με τον ΝΑΤΟ, ο δεν πυροβολούμε ένα τον άλλον. Ή είναι επιτυχία εάν συλλάβουμε όσο δυνατόν περισσότερους πειρατές και βυθίσουμε τα σκάφη τους ή είναι επιτυχία εάν έχουμε ακόμη λιγότερους να αντιμετωπίσουμε λόγω της αποτροπής μας. Εάν επίσης ήταν δική σας η απόφαση πόσο μεγάλη θα θέλατε να είναι η δύναμη, πόσα πλοία και πόσα μέσα θα χρειαζόσασταν κατόπιν κατά την άποψή σας τι πρέπει να γίνει στην ξηρά έτσι ώστε ο κίνδυνος, η απειλή των πειρατών να εξαφανιστεί μονίμως ή να μειωθεί. Ε, κατόπιν ένα ερώτημα από άλλη σκοπιά από τον συνάδελφο Καντέκ που ανέφερε μόλις την αλληλεία. Παρά την απειλή υπάρχει εκεί πέρα εμπορική, εμπορική αλληλεία και το ερώτημα το οποίο εγώ θέλω να θέσω από μια άλλη κατεύθυνση, εμείς στο πλαίσιο της επιχείρησης αυτής είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε, να υποστηρίξουμε τους Ομαλούς αλληλείς που ίσως θέλουν εκεί να πιάσουν κάνα ψάρι. Έτσι ώστε Ε, γιατί οι εμπορικοί στόλοι εκεί πέρα οι υπόλοιποι έχουν αδειάσει τελείω τη θάλασσα και αναγκάζονται αυτοί οι άνθρωποι να αντιδράσουν θετικά στην πρόσκληση, αν θέλετε, να γίνουν πειρατέ εφόσον δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν. Θα μπορούσαμε να εγγυηθούμε αυτή την εμπορική ζώνη 210 μιλίων. Η Σομαλία προφανώς δεν μπορεί να το κάνει από μόνη της. Προστατεύουμε και τους Σομαλούς ψαράδες που θέλουν να ψαρέσουν, να ψαρέψουν και να μπορέσουν έτσι να βγάλουν το ψωμί τους. Και νομίζω καλύτερο θα ήταν να γίνει αυτό συστηματικά έτσι ώστε να γίνουν και λιγότεροι άνθρωποι πειρατές και οι ψαράδες να ξαναγυρίσουν στο ψάρεμα. Ο κύριος Γιάννης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή λόγω τη σοβαρότητα του θέματο, αλλά είναι πολύ δύσκολο να είναι κανεί συνοπτικό και σύντομο. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον υπονάβαρχο Χάτσον για τι πληροφορίε που μα έδωσε και συμφωνώ με αυτού που είπαν ότι πρέπει οπωσδήποτε να διαβιβάσετε αυτά τα συγχαρητήρια σε όλου αυτού οι οποίοι είναι τα πληρώματα των πλοίων τη Αταλάντα που εργάζονται επί οποίο στην επιχείρηση αυτή. Δεν είναι περιττό να τονίσουμε ότι αυτή η ανάπτυξη ναυτικών δυνάμεων, άλλων ναυτικών καλύτερα δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πολύ σημαντική. Είναι κάτι το οποίο δεν είχε γίνει ποτέ στο παρελθόν, από τότε που ξεκίνησε η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι επίσης πολύ σημαντική περιοχή διέλευσης, ένα εμπορικό σταυροδρόμιο, ο κόλπος του Άντεν και η περιοχή της Σομαλίας, μια πολύ μεγάλη σημασία και επομένως είναι απαραίτητο να υπάρχει μια ανάπτυξη δυνάμεων στην περιοχή αυτή. στο 11 μήνες του 2009 ήδη η επιχείρηση Αταλάντα επέτυχε σημαντικούς στόχους. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε κύριε Ναύαρχε πόσες πράξεις πειρατείας έγιναν το 2007, 2008 και 2009. Και στη συνέχεια θα ήταν χρήσιμο να γνωρίσουμε και ποιο είναι το συνολικό κόστος αυτής της επιχείρησης ή τουλάχιστον το κόστος το οποίο επομίστηκε η επιχείρηση αυτή μέσα στους τελευταίους 11 μήνες. Είναι φυσικά μια ενέργεια η οποία βασίζεται σε ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και είχαν σαν στόχο να εξασφαλίσουν τη λειτουργία του σχεδίου για την ε, ε, διατροφή του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής της ε, Σομαλίας από τα Ηνωμένα Έθνη. Η Ισπανία προφανώς ενδιαφέρεται ιδιαίτερα και γι' αυτό η Αταλάντα ήταν μια γαλλο-ισπανική πρωτοβουλία καταρχήν. Η Ισπανία ενδιαφέρεται όχι μόνο για τα θέματα τα αλλιευτικά, αλλά επειδή τώρα έχουμε μεγαλύτερη ευαισθησία για το θέμα του μικρού Αλακράνα, ο οποίος έχει συλληφθεί και κρατείται όμοιρος. Όπως ξέρετε, συνελήφθη μαζί με άλλους 30 που ήταν το πλήρωμα ενός ισπανικού πλοίου. Νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση υπήρξε τεράστιος αντίκτυπος στα μέσα ενημέρωσης και είναι προφανές ότι Προφανώς δεν μπορούν τα μέσα ενημέρωσης να καθορίσουν τους στόχους μιας επιχείρησης, αλλά υπάρχει μια πολύ μεγάλη ευαισθησία στο θέμα αυτό αλλά είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη και η προστασία των ατόμων αυτών που είναι όμοιροι και γι' αυτό το λόγο να δράσουμε με προσεκτικό και σόφρονα τρόπο. <clears throat> και γι' αυτό, καταλήγω να σας πω κύριε Νάβαρχε αν οι χώρες οι οποίες συμμετέχουν στην Αταλάντα έχουν εξετάσει να υπάρξει και μια επέκταση της περιοχής προστασίας προς τα νότια. Είναι φανερό ότι τα μικρά αυτά σκάφη που βρίσκονται μακριά από τη ζώνη προστασίας θέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο και το έκαναν φυσικά εν γνώση τους. Αλλά θα ήταν χρήσιμο να ξέρουμε να γνωρίζουν οι εφοπλιστές και οι πλοίαρχοι των πλοίων τι ακριβώς κινδύνους διατρέχουν εάν περάσουν σε αυτές τις ζώνες. Τώρα φυσικά εμείς θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και την ε, ε, ελευθέρωση του πληρώματος του αλληλευτικού πλοίου στο οποίο βρέθηκε και αυτό το, αυτός ο νέος και να υπάρχει και καλύτερη προστασία των αλληλευτικών πλοίων. Είπε ο ο Ροσκάντεκ ότι η Γαλλία χρησιμοποιεί πια τώρα στρατιωτικές, τακτικές στρατιωτικές μονάδες στα αλληλευτικά πλοία. Στην Ισπανία αυτό δεν επιτρέπεται από την τρέχουσα ισπανική νομοθεσία και επομένως η Ισπανία ζήτησε από τους ε, εφοπλιστές να έχουν ιδιωτικές δυνάμεις ασφαλείας. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η δική σας άποψη για το θέμα αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω σε ποιο βαθμό συνεργάζεται η Blackwater με την Ισπανία σε συγκεκριμένο επίπεδο στα, και συγκεκριμένα στο θέμα της, ε, της ε, απελευθέρωσης των ναυτικών του Αλακράνα. Merci, Monsieur et ensuite je laisserai la... και μετά θα απαντήσει στην πρώτη φέτα ερωτήσεων ο Ναύαρχος Χάτσον. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ, κύριε Υπονάβαρχε. Εγώ θα ήθελα να θέσω κάποιες ερωτήσεις επιπλέον, πέρα από τις που μας δώσατε. Πρώτα απ' όλα, στο κέρας Αφρικής, εδώ και καιρό, Έχουμε δυνάμεις ε, του ΝΑΤΟ από την επιχείρηση Enduring Freedom για την καταπολέμηση της ε, τρομοκρατίας, για άλλο λόγο. Υπάρχει εκεί πέρα κάποια μορφή συνεργασίας, ε, ανταλλαγής πληροφοριών ή οποιασδήποτε άλλη συνεργασίας μεταξύ των μονάδων εκείνων της επιχείρησης Enduring Freedom και της επιχείρησης Αταλάντα. Δεύτερη ερώτηση. Ε, όπως είπε και ο κύριος Γκάλερ, έθεσε το ζήτημα της συνεργασίας μεταξύ της Αταλάντας και του ΝΑΤΟ και των ήπα και των λοιπών μονάδων που επιχειρούν στην περιοχή. Υπάρχει μία μονιμοποιημένη δομή της συνεργασίας ή είναι μία συνεργασία ad hoc. Και η συνεργασία αυτή είχε οδηγήσει σε κάποιες ε, συγκρούσεις με πιθανώς άλλους ε, συμμετέχοντες. Τρίτον, είναι νομίζω φανερό πως δεν μπορεί να σταθεί μόνη της η επιχείρηση Αταλάντα, αλλά χρειάζεται μια συνολική πολιτική για την περιοχή. Το ερώτημα λοιπόν, κύριε Υπονάβαρχη, είναι το εξής. Στο πλαίσιο αυτό μια συνολικής ε, πολιτικής. Ε. Η πρόταση της 12ης Νοεμβρίου του Ισπανού Υπουργού Άμυνας είναι θετική. Η πρόταση αυτή ήταν η Αταλάντα να έχει την αποστολή δηλαδή να αποκλείσει την Σομαλική ακτή. Κατόπιν, ένα ερώτημα μετά από αυτά τα οποία είπε ο κύριος ε, Καντέκο, πρόεδρος της Επιτροπής Αλληλείας. Αυτό το οποίο προτείνει ο κύριος Καντέκ, δηλαδή οι δυνάμεις που έχετε στην διάθεσή σας επαρκούν για την αποστολή σας ή χρειάζονται κι άλλες. Και κατά την άποψή σας, μήπως θα ήταν καλύτερο σε αυτή τη σύγκρουση οι Ευρωπαίοι να είναι πιο συγκρατημένοι και να μην αδειάσουν τελείω την περιοχή από ψάρια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ναύαρχη, έχετε το λόγο. Λοιπόν, να απαντήσω. Έχω κάποιες απαντήσεις. Λοιπόν, για αυτό το οποίο με ρώτησε ο πρόεδρος για το τι βλέπουμε στο ευρύτερο πλαίσιο με την πειρατεία. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως υπάρχουν τεράστιες χρηματικές ροές από τις ε, δραστηριότητες πειρατείας. Δεκάδες εκατομμύρια δολαρίων το τελευταίο έτος. Και παρά τον νεοπλουτισμό κάποιων πειρατών με τα σπίτια τους και τα τζίπ εκεί πέρα, το να βρούμε που πάνε τα χρήματα είναι σημαντικό. Αυτό είναι σημαντικό, έχετε ακούσει και τα σχόλια της Υπουργού Εξωτερικών Κλίντον ε, τον Απρίλιο φέτος και στην περίπτωσή μας και η ασφάλεια της Μεγάλης Βρετανίας και λοιπές ε, υπηρεσίες λαμβάνουν ε, πληροφορίε από εμά, αλλά δεν είναι ακριβώς η αρμοδιότητά μου. Θα σας παρέπεμπα σε αυτές τις υπηρεσίες μάλλον κατά πολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Όπως σας είπα, είναι πολύ έξυπνοι αυτοί οι άνθρωποι, είναι επιχειρηματίε θα έλεγα, προσαρμόζονται και για να αναφερθώ λίγο και στα ερωτήματα της αλληλείας, τη μία στιγμή μπορούν να είναι κανονικά νόμιμοι Σομαλοί αλληλείς, ε, έχουν τα δίχτυα τους με τις μεγάλες βάρκες, με τα μικρά βαρκάκια από πίσω, απλώνουν τα δίχτυα και όταν δουν ένα σκάφος και θεωρούν ότι είναι ευκαιρία λένε ας κάνουμε και το ρεσάλτο. Οπότε, ε, όπως σας είπα, έχουν τώρα περάσει στην ε, εμπορία ανθρώπων. Υπολογίζει η πατιαρμοστία του ΟΗΕ 24.000 άτομα ότι έχουν μεταβάσει στην ε, Αραβική Χερσόνησο και χρεώνουν γύρω στα 150 δολάρια το κεφάλι. Οπότε δεν είναι ένα σκληρός πυρήνα πειρατών μπορούμε να στοχεύσουμε, είναι ένα ευρύ φάσμα εγκληματικών δραστηριοτήτων τώρα να αναφερθώ σε κάποια από τα σημαντικά σημεία που ανέφερε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως εάν όλα τα πλοία που πλέον στην περιοχή έρχονταν σε επαφή με το δικό μας το κέντρο ή με το κέντρο στο Ντουμπάι και λοιπούς οργανισμούς ε, υπάρχουν και στο Μπαχρέιν και αλλού στην Άπο Ανατολή ανάλογα κέντρα και ακολουθούσαν αυτές τις ε, συμβουλές δεν θα ήταν σε τέτοιο κίνδυνο. Εμείς υπολογίζουμε ότι γύρω στο 35 με 40% των σκαφών που διαπλέουν την περιοχή δεν ε, έχουν πλήρη ενημέρωση και προσπαθούμε να το βελτιώσουμε αυτό. Συνεργαζόμαστε με τους Αιγυπτίους να δούμε τι θα κάνουμε στο Σουέζ όταν πηγαίνουν νότια, όταν περνάνε τους Σουέζ και κατεβαίνουν νότια. Έχουμε ε, σύνταξη χιλιάδες χάρτες με τους διάβλους που συνιστούμε, τα μέτρα προστασίας, τα έχουμε μοιράσει σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα κέντρα ναυτιλωμένων, ναυτιλιακές εταιρείες, παντού εργαζόμαστε. Αλλά κάποιες από αυτές τις εταιρείες είναι... Έχουν μόνο ένα πλοίο, τους ανησυχεί το κόστος του να λάβουν τέτοια μέτρα, αλλά είναι ανασφάλιστες. Οπότε πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια όσον αφορά δε τις συμβουλές είναι προς όλους τους ναυτιλωμένους και σε όσους έχουν σκάφη αναψυχής και στα αλληλευτικά σκάφη. Και δίνουμε και συγκεκριμένες οδηγίες και σε αυτούς και στους αλληλείς και τους λέμε ότι τα πλοία τα οποία είναι αργοκίνητα, ε, είναι χαμηλά η ίσαλος γραμμή και όλα αυτά, να προσέχουν. Γιατί υπάρχουν και επιθέσεις ευκαιρίας. Οπότε, το πολύ σημαντικό ζήτημα τώρα των ε, Ισπανών και Γάλλων ε, αλλιέων και πώς ε, συντονιζόμαστε. Νομίζω πως έχουμε αρκετά καλές επαφές με το σύνδεσμο των Ισπανών αλλιέων. Υπάρχει εκπρόσωπός του στο επιτελείο μου και με τους Γάλλους συναδέλφους τους, με τις εταιρείες υπάρχει καθημερινή ροή πληροφοριών και με τις δύο οργανώσεις όταν υπάρχει ύποπτη δραστηριότητα. Ε, όπως σα είπα έχουμε αναπτύξει ε, βέλτιστες πρακτικές για αυτά τα σκάφη. Έχω τοποθετήσει εγώ σκάφη ναυτική, αεροσκάφη ναυτική συνεργασία στι Αιχέλες και στη Μομπάσα για να καλυφθεί ολόκληρη η περιοχή. Οπότε νομίζω υπάρχει αρκετά καλή σύνδεση, αλλά μιλάμε για στόλους που είναι διασπαρμένοι σε εκατοντάδε μίλια ωκεανού, για την Δέα Λακράνα ήταν ε, ε, σε ένα σκάφος μεμονωμένο και με τις δυνάμεις βεβαίως που έχω στη διάθεσή μου δεν μπορώ να συνοδεύσω το κάθε πλοίο ξεχωριστά. Οπότε κάνουμε ό,τι μπορούμε, δίνουμε πληροφορίες ε, και στις δύο ενώσεις αλλιέων και το άλλο θέμα το οποίο αναφέρθηκε είναι πώς θα διασφαλίσουμε συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μαχικών Δυνάμεων στον Μπαχρέιν, του ΝΑΤΟ, για να έχουμε μία μόνιμη παρουσία. Η συνεργασία αυτή περνάει από το ΣΕΙΔ, το Κοινό Κέντρο Πρόληψης ε, Συγκρούσεων. Έχουμε μία σύσκεψη κάθε μήνα στο Μπαχρέιν. Είναι συμπρόεδρος η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε 22 χώρες και οργανισμούς που συμμετέχουν από την Ινδία, Κίνα, Ρωσία και το δικό μου το επιτελείο και ένα κέντρο του Ηνωμένου Βασιλείου στο Μπαχρέιν, καθώς και συγκεκριμένες στοιχείες βεβαίως της ε, καταπολέμησης πειρατείας. Είναι ένα φόρουμ, δεν έχει ε, αρμοδιότητες εκτελεστικές όσον αφορά τι επιχειρήσει. Απλά μοιραζόμαστε σχέδια, συντονιζόμαστε για να μην είμαστε όλοι μαζί δίπλα-δίπλα στην Σαλάλα ή όλοι μαζί στην Μομπάσα, να υπάρχει μια διασπορά σε ολόκληρη την λεκάνη της Ομαλίας ε, και τον κόλπο του Άντεν για να υπάρχει και παρουσία συνεχής ε, στον ε, διάβλο. Επίσης, ε, τα αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας συντονίζονται. Οπότε ο συντονισμός μας στο θέατρο των επιχειρήσεων είναι πολύ καλός και ως Ευρωπαϊκή Ένωση ΝΑΤΟ και ως Ευρωπαϊκή Ένωση Κέντρο Ναυτικής Ασφάλειας. Όπως ακούσατε, εμείς επικεντρωνόμαστε στο πρόγραμμα επισητισμού, στη βοήθεια της Αφρικανικής Ένωσης και στην ναυτιλία και την καταπολέμηση των πειρατών. Το ΔΕ άλλο κέντρο ασφάλειας τη ναυτιλία ε, έχει σχέση βεβαίως με την επιχείρηση Enduring Freedom, αλλά οι δυνάμει που έχουν στον Ινδικό ωκεανό έρχονται σε συνεννόηση μαζί μας. Οπότε νομίζω η γενική εικόνα είναι πολύ καλή. Οπότε λειτουργεί αυτό το κέντρο το Τώρα, η άλλη ερώτηση που μου κάνατε πόσα πλοία χρειαζόμαστε. Ε, κανένας ναύαρχος δεν θα σας πει αυτά που έχω μου φτάνουν. Πάντα χρειαζόμαστε περισσότερα. Έχουμε 2 εκατομμύρια τετραγωνικά μίλια περιοχής. Δεν καλύπτονται με 6 ε, πλοία αποτελεσματικά και να μπορούμε να διαβεβαιώσουμε το εμπορικό ναυτικό ή τους ψαράδες ότι δεν θα υπάρχει πειρατεία. Οπότε Πρέπει να υπάρχει σταθερή υποστήριξη από τα κράτη-μέλη. Εγώ συνεργάζομαι αποτελεσματικά με τη Στρατιωτική Επιτροπή και του εκπροσώπους όλων των κρατών μελών για να βρούμε μια ρεαλιστική λύση, γιατί υπάρχουν και άλλε ανάγκε και τι ξέρουμε όλοι ε, που πρέπει να καλύψουν οι ενοπλέ δυνάμει μα. Οπότε έχουμε ένα αρκετά καλό πακέτο θα έλεγα. Κάποιο ρώτησε για μέτρο αποτελεσματικότητα, με τι μετράμε την επιτυχία μα ή μήπως κάνουμε απλά βόλτε θάλασσα. Ξέρω πώ είμαστε αποτελεσματικοί γιατί μιλάω με του ανθρώπου που περνάνε από την περιοχή. Τα πλοία, οι ασφαλιστικέ εταιρείε, οι ενώσει εφοπλιστών, όλοι όσοι κινούνται εκεί καθημερινά και βεβαίω οι αλλοί ε, τόνου και λοιποί, είτε μιλάμε για διεθνή αναγνώριση του διάβλου, των ε, ενεργειών μας, των διαδικασιών μας, των οδηγιών που δίνουμε, υπάρχει διαφορά. Το ποσοστό επιτυχίας ειδικά στον κόλπο του Άντεν από το να κάνει επίθεση και να καταλάβει ένα πλοίο πειρατής, ε, αυτές οι περιπτώσεις μειώνονται συνεχώς. Βεβαίως, όπως σας είπα, η περιοχή είναι τεράστια, η απόσταση μας είναι κάτι το οποίο μας ε, βασανίζει και έχει και κόστος η επιχείρηση. Τα κράτη-μέλη ε, πληρώνουν βεβαίως το κόστος των σκαφών και αεροσκαφών με τον προπολογισμό του. Έχουμε εμεί ένα μικρό προπολογισμό γύρω στα 9 εκατομμύρια ευρώ για το επιτελείο, για όλη την υποδομή, επικοινωνίε, τον ιστοσελίδα που ανέφερα, τη σύνδεση δηλαδή. Οπότε είναι μικρό αυτό ο κεντρικό προπολογισμό. Η πλειοψηφία του κόστου είναι στα κρατημέλη. Τώρα, θα παίξει ρόλο εάν κάνουμε μεγαλύτερη την περιοχή ευθύνη. Είναι κάτι που συζητάμε με τον Διεθνή Οργανισμό Αφιλία και τι ναυτιλιακέ εταιρείε τακτικά και αυτό το οποίο λέμε συνεχώ είναι ε, να προσέχουμε στην αφιλία και παρά το ότι δύο πλοία κατελήφθησαν εκτός αυτής τη περιοχής, τα περισσότερα καταλαμβάνονται από του πειρατέ εντό αυτή τη περιοχή. Οπότε πριν διευρύνουμε την περιοχή ε, ευθύνης, καλά θα κάνουμε να δούμε το τι γίνεται στην περιοχή που καλύπτουμε τώρα. Τέλος, για αγήματα προστασίας ε, εμπορικών πλοίων. Πρώτα απ' όλα για το πρόγραμμα ε, επισητισμού του ΟΗΕ. Εγώ ευχαρίστως να βάλω 12 πεζοναύτες, ειδικέ δυνάμεις, οτιδήποτε, σε ένα πλοίο και μετά έρθουν οι πειρατές αλλά θέλει πάρα πολλές εγκρίσεις από το κράτος σημαίας, από το κράτος σημαίας του, ε, της χώρας που θα δώσει το άγημα, μετά θέλει κανόνες εμπλοκής, είναι δύσκολα τα πράγματα. Και όπως είπα, όταν τα πλοία αυτά έχουν σημαία Κομόρας, Marshall Islands, Βόρειας Κορέας, είναι δύσκολα. Αλλά προσπαθούμε. Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, ένα πλοίο το οποίο θεωρείται ευάλωτο. Ε, είναι πολύ πιο εύκολο για μένα να βάλω εκεί πέρα ένα άγημα. Και έχει συμβεί αυτό γιατί είναι εύκολη η διαδικασία εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι δική μας ε, οι άνθρωποι και τα σκάφη, οπότε μπορούμε να ε, έχουμε επαρκή προστασία. Τι γίνεται τώρα με την Ισπανία και την Γαλλία και τα αλληλευτικά του σκάφη, αν είναι δηλαδή στρατεύματα ή ιδιωτικέ ε, δυνάμει. Αυτό είναι θέμα των εθνικών αρχών. Έχουμε δει το τι κάνει η Αμερική και το τι έγινε μετά την επίθεση στο Μέρ Καλαμπάμα. Και εκεί πέρα πολεμικά πλοία τον είπα συνόδευαν. Οπότε εξαρτάται με το τι κάνει κάθε χώρα το αντιμετωπίζει διαφορετικά. Και εμείς συμπληρώνουμε και υποστηρίζουμε τις δύσκολες αυτές αποφάσεις, ειδικά όταν ε, επιχειρούν σε μια τέτοια περιοχή. Ελπίζω να κάλυψα όλες τις ερωτήσεις σας. Ε, εάν όχι, να επανέλθω κύριε Πρόεδρε. Ναι, ναι, οι Σομαλοί ψαράδες. Υπάρχει ένα ζήτημα πράγματι. Αυτοί οι άνθρωποι είναι μεροδούλοι μεροφάοι ψαρεύουν κοντά στην ακτή. Η πλειοψηφία των ε, σκαφών ε, δε αυτών ε, ψαρεύουν σε μια αποκλειστική οικονομική ζώνη την οποία ακόμη δεν έχει διεκδικήσει η Σομαλία και τα περισσότερα από αυτά τα σκάφη είναι από μέρη όπως η Εμένη. δεν είναι μεγάλα αλληλευτικά σκάφη και με διαβεβαιώνουν τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη πως τα ευρωπαϊκά ληστικά σκάφη είναι έξω από τα 200 μίλια. Οπότε τα παρακολουθούμε, ξέρουμε που βρίσκονται. Το παρακολουθούμε στο κοινό κέντρο επιχειρήσεων. Οπότε εντός της ζώνης των 200 και των 12 μιλίων δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη αλληλεία, η σομαλική δηλαδή, είναι απλά για επιβίωση και δεν έχω δει κανένα μεγάλο στόλο, είτε μιλάμε σαουδαραβικό είτε ιεμενικό. Ε, το τι συνέβη στο παρελθόν τώρα δεν μπορώ εγώ να το σχολιάσω. Δύο ερωτήματα για την ΟΗΕΦ και για την πρώτη. Η επιχείρηση μόνιμη ειρήνη, Ensuring Freedom, την, ε, την ε, κάνουν οι Αμερικανοί με, δι, με τις δυνάμεις αυτές οι οποίες προέρχονται από τον Μπαχρέν. Είναι η 151 και η 450. Η μία από τις δύο μονάδες ασχολείται με την αντιμετώπιση της πειρατείας και η άλλη με το ευρύτερο θέμα ασφαλείας στην περιοχή. Επειδή κάνουμε αυτές τις συναντήσεις μας στον Μπαχρέν για να υπάρξει καλύτερα συντονισμός, επειδή οι τρεις δυνάμεις, η CMF, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθούν να έχουν μια κοινή προσέγγιση και δεν μας δεσμεύει κάτι ανά της Κίνας και της Ρωσίας. Προσπαθούμε να έχουμε λοιπόν ένα συντονισμό και τα στοιχεία της κοινή αυτής δύναμης που αντιμετωπίζει την πειρατεία θεωρούμε ότι πρέπει να είναι αντικείμενο συνεργασίας. Τα ευρύτερα θέματα τα αντιμετωπίζουμε χωριστά βέβαια, από την, από την ομάδα αυτή που βρίσκεται στο Μπαχρέιν και αυτά είναι τα ωφέλη τα οποία μπορούν να αποκομίσουν μεγάλοι φορείς σαν την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, το CMF σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Και υπάρχουν βέβαια ανεξάρτητες δυνάμεις όπως η Ιαπωνία, η Κίνα, η Μαλαισία που μπορούν όμως να συνεργάζονται μαζί μας για το καλύτερο αποτέλεσμα. Νομίζω ότι έτσι έχω απαντήσει το ερώτημά σας. Ευχαριστώ κύριε Ναύαρχε. Μια δεύτερη φέτα ερωτήσεων, τέσσερα, τεσσάρων ερωτήσεων, κύριος Έλεα. Κύριε Ναύαρχε, α, είσαμε ως ε, πολιτικοί πως ε, τονίσατε τη σχέση σαφίους ε, πολιτικής αποστολής και στρατιωτικής επιτυχίας. Και έχω ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Στα ΜΜΕ αναφέρθηκε μία περίπτωση μιας γερμανικής φρεγάτας η οποία συνέλαβε πειρατές ε, ανοιχτά της ε, Σομαλίας και στο περιστατικό αυτό σκοτώθηκε και ένας πειρατής και μετά αναρωτιόντουσαν στην γερμανική κυβέρνηση και στο Ευρωπαϊκό Επιταλείο κατά πόσο μπορούν να τους παραδώσουν στην Κένια. Και αποφάσισαν να μην τους παραδώσουν στην Κένια αλλά να τους αφήσουν πάλι ελεύθερους. πόσο σαφείς είναι οι κανόνες, πότε εκδίδεται κάποιος και πότε όχι και δεν καταλήγει σε δικαστήριο ή όχι. Και δεύτερο ερώτημα, πληροφορηθήκαμε από τα ΜΜΕ πως ε, ο βαθμός της οργάνωσης της πειρατείας στη Σομαλία έχει περάσει σε άλλα επίπεδα. Μιλάμε για στρατιωτικές ε, πληροφορίες πλέον και μυστικές υπηρεσίε θα λέγαμε που έχουν πολύ σοβαρές γνώσεις για την κίνηση της εμπορικής ναυτιλίας. Πώς το αντιμετωπίζετε αυτό, συνεργάζεστε με πολιτικές αρχές, ποιες πληροφορίες έχετε εσείς για τη νέα αυτή κατάσταση και για τις μεγαλύτερες δυνατότητες απόκτησης ε, πληροφοριών των πειρατών. Και τέλος, Μιλήσατε για επιτυχία, δεν το αμφισβητεί κανείς, εγώ σας συγχαίρω βεβαίως, αλλά ποια είναι η εκτίμησή σας. Η επιτυχία όταν θα φύγει από εκεί η ευρωπαϊκή δύναμη θα συνεχιστεί ή θα επανεμφανιστεί η πειρατεία και έχουμε επιτυχία μόνο όσο είναι ε, μόνιμη εκεί πέρα η στρατιωτική παρουσία. Κύριε Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Ναβαρχέ για τις εξηγήσεις που μας δώσατε. Και εγώ ως Ισπανής πρέπει να πω ότι ανησυχούμε πάρα πολύ για τα τεκτενόμενα, για τους οικείους των ανθρώπων οι οποίοι έχουν συλληφθεί και κρατούνται όμοιροι παραγωγή χάρη. Έχουμε ένα πρόβλημα. Αλλά είπατε ότι δούλεψε καλά η Αταλάντη. Η Αταλάντα μάλλον. Αλλά θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Βέβαια. Υπάρχει μια μείωση του αριθμού των ομήρων, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά επεισόδια, γιατί οι πειρατές εξυγχρονίστηκαν έχουν προσαρμοστεί στις νέες τεχνολογίες, στους νέους τρόπους σύλληψης πλοίων, πολύ πιο γρήγορα από εμά. Η συμφωνία που είχε συναυθεί πέρσι παρατάθηκε η ισχύ της, αυτή είναι μια καλή συμφωνία, αλλά θα πρέπει να την ενημερώσουμε το ταχύτερο δυνατό που μας επιτρέπουν οι συγκυρίες. <clears throat> Έχω λοιπόν δύο ερωτήματα τα οποία θα αναθέσω από αλλιευτική άποψη, γιατί και εγώ είμαι μέλος της Επιτροπής Αλλιείας και θεωρώ ότι είναι θεμελιώδη ερωτήματα αυτά. Καταρχήν, η διεύρυνση της περιοχής προστασίας. Η, η συμφωνία λέει προστασία ευαλώτων πλοίων που πλέουν στις ακτές της Σομαλίας. Τώρα, είναι τεράστια η ακτογραμμή της Σομαλίας, αλλά είναι μικρή αυτή η περιοχή. Και εξάλλου τα αλληλευτικά πλοία είναι η προτεραιότητα των πειρατών αυτή τη στιγμή. Επομένω, τα αλληλευτικά σκάφη είναι, δεν είναι ένα ακόμα ευάλωτο είδο πλοίων. Είναι τα πιο ευάλωτα πλοία γιατί είναι αυτά τα οποία πληρώνουν τα περισσότερα λίτρα. Δεν έχω γνωρίσει ποτέ έναν άβαρχο που να λέει ότι έχει πάρα πολλούς πόρους και δεν χρειάζεται παραπάνω. Πάντα ζητάτε περισσότερο, αλλά όταν ζητάτε να έχετε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, χρειάζεται πράγματι να υπάρχει μια διεύρυνση της περιοχής προστασίας. Και αν υπάρξει αυτή η επέκταση της προστασίας για τα αλληλευτικά πλοία, Μήπως <clears throat> αυτό θα έχει κάποιο αποτέλεσμα. Η Ισπανία ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την Αταλάντα, λοιπόν, όχι μόνο οι πειρατές. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Λιζέκ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, δύο ζητήματα θα ήθελα να θέσω. Το πρώτο ερώτημα προκύπτει από αυτό που είπε ο κύριος Έλε. Πρώτον, πώς αξιολογείται τον εξοπλισμό των πειρατών. Επίσης πώς νομίζετε ότι θα εξελιχθεί, θα αυξηθεί, θα μειωθεί, θα υπάρξουν αλλαγές γιατί κάποιος είπε ότι έχει, έχουν μειωθεί οι επιχειρήσεις των πειρατών. Αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένω κάποια στιγμή θα σταματήσουν. Και ένα ακόμα ερώτημα. Ενδεχομένω ε, δεν θα έπρεπε να το ρωτάω σε εσά, ενδεχομένω σε κάποιον πολιτικό να έπρεπε να απευθύνω το ερώτημα. είναι σαν ε, να θεραπεύουμε σε ιατρικού όρου τα συμπτώματα αντί τους λόγους ε, μια ασθένεια. Μήπω θα μπορούσατε να μα πείτε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να εξαλειφθεί το πρόβλημα, η ασθένεια αυτή της πειρατείας. Γιατί νομίζω ότι σε τελική ανάλυση κάτι θα πρέπει να κάνουμε ε, και θα υποχρεωθούμε να απαγορεύσουμε τα πλοία μας στην περιοχή. Διαφορετικά δεν βλέπω πώς μπορούμε να διατηρούμε τους στόλους μας σε μια τόσο επικίνδυνη κατάσταση. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε για να μπορέσει να εξαλειφθεί το πρόβλημα. Ευχαριστώ Άντι Νάβαρχε και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την ε, δέσμευσή σας και εκφράζω την ικανοποίησή μου για τα αποτελέσματα της επιχείρησης αυτής της αποστολής Αταλάντα. Θα ήθελα εδώ τώρα να εμβαθύνω, εμβαθύνω μάλλον, λίγο περισσότερο αυτά που αναφέρατε σε σχέση με την τροποποίηση του πειρατικού φαινομένου της ε, παρανομίας που σοβεί στις θάλασσες της Σομαλίας που είναι μια ευρεία γεωγραφική περιοχή. Έχετε λοιπόν το φαινόμενο ότι μετατοπίζεται προς τα νότια η πειρατική δραστηριότητα και επίσης ότι αλλάζει και η φύση της, η φύση αυτών των φαινομένων. Δηλαδή ότι κυρίως ασχολούνται με το ε, λειτουργήμα της εμπορίας ανθρώπων. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω αν αυτό συνδέεται με άλλες εγκληματικές ενέργειες και σε ό,τι αφορά την ε, λαθρεμπορία ανθρωπίνων όντων, ποιες είναι οι μορφές αυτής της, μετα... αυτής της ροής λαθρεμπορίας, από πού έρχονται και πού πηγαίνουν. Ένα δεύτερο ερώτημα που θέλω να θέσω θα ήθελα να καταλάβω καλύτερα ποια είναι η δική σας άποψη σε σχέση με τις αιτίε αυτού του φαινομένου, δηλαδή της τροποποίησης της δραστηριότητας των πειρατών. Θα μπορούσε κανείς να αποδώσει αυτή την άλλαγη στην αποτελεσματικότητα της επιχείρησης Αταλάντα και άλλων αντίστοιχων ενεργειών προστασίας ή οφείλονται κυρίως σε εσωτερικούς λόγους που έχουν να κάνουν με την εσωτερική κατάσταση που επικρατεί στη Σομαλία ή το ευρύτερο περιφερειακό πλαίσιο. Και τέλος, ποια είναι η άποψή σας σε σχέση με τη θεραπεία που μπορεί να δοθεί στα φαινόμενα αυτά, δηλαδή πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε, αν η, η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να αντιμετωπίσει και τέτοια φαινόμενα και νομίζω <clears throat> ότι έχετε εσείς μια επιφυλακτική στάση σε σχέση με μια ενδεχόμενη υπερεπέκταση αυτής της ε, αποστολής που θα εξαντλήσει τις δυνάμεις της αν υπάρχει επέκταση σε μεγαλύτερο γεωγραφικό τρόμο, μήπως, τρό, χώρο. Μήπως λοιπόν μπορεί η αποστολή αυτή να αντιμετωπίσει και τα θέματα ανθρωπίνων αλλά θεμπορίες ανθρωπίνων όντων ή αυτό θα εξαντλήσει τις δυνάμεις της. Υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει μια πιο άμεση λοιπόν εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σομαλία, ίσως με μια συγκεκριμένη δράση της ε, ε, πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Η κυρία Ευχαριστώ πολύ. Δύο ερωτήματα ήθελα να θέσω, αλλά μία ήδη ετέθη όσον αφορά την ε, κατάρτιση των ε, δυνάμεων ασφαλείας. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να διερευνηθεί το θέμα θα ήθελα να μου πείτε περισσότερο, περισσότερα πράγματα για τους λόγους. Και μία ακόμη ερώτηση για τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αρχών της Δημοκρατίας των Σεχελών για τη μεταφορά των ε, πειρατών ε, στη χώρα τους. Ε, μέχρι τώρα, μέχρι τώρα στην Κένια τους μεταφέρουμε, μέχρι να δικαστούν. θα, υπάρχουν, ε, θα υπάρξει κοινοτική νομική εμπειρογνωμοσύνη. Ελπίζω ότι σύντομα θα υπογραφούν οι σχετικές συμφωνίες. Κατά τη γνώμη μου είναι ένα θετικό βήμα, αλλά πώς θα εξασφαλίσουμε την, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στις ΣΕΙΧΕΛΕΣ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ναύαρχη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την δεύτερη σειρά τόσο σημαντικών και χρησίμων ερωτήσεων. Το θέμα του διεθνούς δικαίου είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα τα οποία θέσατε και ακούσαμε γι' αυτό το επεισόδιο για την γερμανική φρεγάτα και τη δυνατότητα δίωξης κατά των πειρατών. Τίποτα δεν με ματαιώνει περισσότερο ή και τους ναύτες μου, ακόμα και τα πλοία μου, όταν είμαστε λίγα μίλια έξω από τις ακτές των, ε, της Σομαλίας και βλέπουμε ότι έρχονται άτομα γεμάτα ενόπλα άτομα, τα οποία δεν κάνουν απολύτως τίποτα εκείνη τη στιγμή, αλλά ουσιαστικά συνομωτούν να κάνουν στο άμεσο μέλλον μια πειρατική ενέργεια που είναι ένα αδίκημα βάσει του δικαίου της θάλασσας και της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών. Βέβαια, κανένα από τα κράτη της Αφρικής δεν έχει ενσωματώσει αυτό στο εθνικό του δίκαιο. Έχουμε συμφωνίες μεταφορά στην Κένια και στις Σεϊχέλες, αλλά θα πρέπει να σεβαστούμε το νομικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν αυτές οι χώρες. Επομένως, συνεργαζόμαστε με τις χώρες αυτές να δούμε και ποια είναι η άποψή τους. Γι' αυτό, κατά καιρόν, αυτή η ύποπτοι για πειρατεία απελευθερώνονται. Και συνεργαζόμαστε με τις αρχές της να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον, αλλά πρέπει να σεβαστούμε και το νομικό τους πλαίσιο. Οι πλευρές ελέγχου λοιπόν και διοίκησης μεταξύ των πειρατών βελτιώνονται όλο και περισσότερο, έχουν μεγαλύτερη συνοχή από ό,τι στο παρελθόν, <clears throat> αλλά υπάρχει και σχέση με τις αρχές οι οποίες εμπλέκονται στο διεθνές με αυτούς οι οποίοι εμπλέκονται στην καταδίωξη του διεθνούς εγκλήματος και με τις ακτές της παράκτης περιοχές για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε τον αγώνα κατά της πειρατείας και πρέπει κοντά στις ακτές της Ομαλίας να έχουμε συνεργασία με όλους αυτούς τους φορείς. Το ερώτημα. Αν μπορούμε να εγγυηθούμε την επιτυχία για το μέλλον. Αν αλλάξει η φύση της δύναμης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιοι ανέφεραν το θέμα της ανοικοδόμησης στην περιοχή αυτή. Βέβαια, οι αιτίε του φαινομένου είναι στην ίδια τη Σομαλία. Αυτό που βλέπουμε τα συμπτώματα. Είναι άτομα τα οποία δεν έχουν τίποτα να χάσουν ουσιαστικά και αποδίδονται και επιδίδονται στην πειρατεία. Χρειάζεται λοιπόν να θέσετε αυτό το ερώτημα σε άτομα τα οποία έχουν περισσότερη γνώση των επιτοπίων θεμάτων από μένα και ο συντονισμό τη υποστήριξη μεταξύ τη Αφρικανική Ένωση, των ΗΠΑ, τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του ΟΗΕ είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει και θα πρέπει αυτό να το αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. <clears throat> Αν είναι επιτυχεί αυτέ οι ενέργειε, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε ίσω να περιμένουμε να υπάρξει και μείωση στι πειρατικέ ενέργειε. Σε ό,τι αφορά τώρα τη διεύρυνση τη περιοχή προστασία, εγώ κατανοώ τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα πλοία τα οποία συλλαμβάνονται εκτό τη περιοχή προστασία και υπήρξαν τέσσερις τέτοιες περιπτώσεις. Το ένα ήταν στη Μασκάτη, ήταν στο, στο Ομάν ουσιαστικά, ήταν πολύ πιο βόρεια. Ένα άλλο στι Σεχέλε, ένα στη Μαδαγασκάρη. Το να μπορέσουμε να, να καλύψουμε μια ευρύτερη περιοχή που θα προστατεύσει περισσότερα πλοία, αυτό σημαίνει περισσότερες ναυτικές δυνάμεις. Αλλά το να έχουμε μια ευρύτερη περιοχή χωρίς να έχουμε τους απαραίτητους πόρους, αυτό δεν αυξάνει το επίπεδο ασφαλείας. Σε ό,τι αφορά τώρα τα αλλιευτικά πλοία τα οποία έχουν συλληφθεί, παρά την ε, πολυπλοκότητα της, περιοχής, της περίπτωσης Αλακράνα, τα άλλα πλοία τα οποία ε, έχουν συλληφθεί το 2008 ήταν εμπορικά πλοία και όχι αλληλευτικά πλοία, εκτός από δύο Αιγυπτιακά τα οποία συνελήφθησαν. Επομένως, το κύριο, κύριο όγκος της πειρατείας αφορά τα εμπορικά πλοία το αν θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις πρακτικές μας. Όπως είπαμε, η λύση βρίσκεται στις ακτές και στο έδαφος της Σομαλίας. Εμείς θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίσουμε πολλές φορές αντικρουόμενες αιτήσει από διάφορες κατευθύνσεις και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε όλη και μεγαλύτερη υποστήριξη είτε στα αληφτικά πλοία είτε στα εμπορικά πλοία που περνούν από την περιοχή αυτή. Σε ό,τι αφορά το, τα αριθμητικά στοιχεία το να αντιμετωπίζουμε τις ιστορικές τάσεις. Ναι, είναι σαφές ότι υπάρχει μια αλλαγή τάσεων. Ο κόλπος του Άντεν μέχρι στιγμής ήταν σχετικά γαλήνιος. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να αποσυρθούμε από εκεί. Αλλά οι πειρατές και αυτοί αλλάζουν τακτικές συνέχεια. Είδαμε στο παρελθόν να πηγαίνουν ορισμένοι στην Ιεμένη <clears throat> και να μεταφέρουν ε, μετανάστες οικονομικούς να γυρίζουν στη συνέχεια με εξοπλισμό στρατιωτικό για πειρατεία, να χτυπάνε ένα πλοίο και μετά να ξαναγυρίζουν στην Ιεμένη να φέρουν άλλου μετανάστε. Δηλαδή έχουμε μια τέτοια αντιμετώπιση που είναι ευέλικτη και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε μια σωστή συνεργασία με την ε, υπατιαρμοστία του ΟΗΕ για τα θέματα των προσφύγων και των μεταναστών, να έχουμε μια καλύτερη συνεργασία με τους Γεμενίτες και τους Σομαλούς, τις αρμόδιες αρχές και φυσικά πρέπει να αντιμετωπίσουμε και ανθρωπιστικού χαρακτήρα καταστάσεις όπου κάποια άτομα αφήνονται στη θάλασσα χωρίς καμιά προστασία στην τύχη τους. Είναι σημαντικό λοιπόν να εξασφαλίσουμε και την ασφάλεια στη θάλασσα. Αλλά η λύση για τα 24.000 άτομα τα οποία θέλουν να φύγουν από τη Σομαλία δεν είναι διαφορετική από αυτούς οι οποίοι θέλουν να πάνε στη Σομαλία. Η ζωή είναι πολύ δύσκολη, επομένω θα πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να ανοικοδομήσουμε την περιοχή αυτή τη Σομαλία και ελπίζω ότι βελτιωθούν οι προσπάθειες των ΗΕ. Συλλογή πληροφοριών. Δεν νομίζω ότι παίρνουν πληροφορίες ευαίσθητες από τη δική μου δύναμη οι πειρατές, αλλά είναι μικρή η... μικρό το εύρος του διάβλου του, του κόλπου του Άδεν. Επομένως, είναι σχετικά εύκολο να ξέρει κανείς πού βρίσκεται το κάθε πλοίο. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητο να έχουμε καλό διάλογο μεταξύ των ε, εμπορικών πλοίων και της δύναμης αυτής της Αταλάντα εν τέλει. Η σύνδεση μεταξύ της Αταλάντας και τις ε, αλλαγές που γίνονται στην ε, περιοχή του Πούντι, ιδίως αλλά και γενικά στη Σομαλία. Εδώ πρέπει να πω ότι η Αταλάντα και οι προσπάθειες που γίνονται από το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ιαπωνία, τον συνασπισμό, όλοι αυτοί δίνουν το μήνυμα ότι υπάρχει πράγματι μία μεγαλύτερη ασφάλεια. Το γεγονός ότι υπήρξε η συμφωνία αυτή με την περιοχή του Πούντ, η οποία έχει συμφωνία να αφήνει τις δυνάμεις μας να ενεργούν στην περιοχή αυτή και το γεγονός ότι το αποδέχεται ότι είναι σημαντικό αυτή η περιοχή, είναι πολύ θετικό. Τελικά, πιστεύω ότι η ύπαρξη μιας μεγαλύτερης αποτροπής θα ελαττώσει εν καιρό την πειρατεία. Για το πού πηγαίνουμε στο μέλλον, και αυτό μπορείτε να το συζητήσετε και πάλι, όταν ε, έχετε τους εκπροσώπους της ε, πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω. Και τώρα ετέθη το ερώτημα γιατί τα εμπορικά πλοία δεν έρχονται σε επαφή μαζί μας. Ούτε και εγώ ξέρω. Ο διάλογος μας με τις μεγάλες εταιρείες δεν εταιρείε σαν τη Merckx, τη Shell, την P&O αυτές καταγράφουν τα πλοία τους. Είναι μικρές εταιρείε οι οποίες δεν το κάνουν αυτό. Υπάρχει το θέμα του κόστους, θεωρώ. ότι θα τους κοστίσει περισσότερο. Είναι το εμπορικό συμφέρον, ότι δεν θέλουν να ξέρουν πού είναι τα πλοία τους οι άλλοι. Είναι επίση και ορισμένοι που λένε ότι αν καταγραφούμε θα μεταδοθούν αυτέ τι πληροφορίε κατευθείαν στου πειρατέ. Θα τηλεγραφηθούν στου πειρατέ. Λοιπόν, Υπάρχουν πολλοί λόγοι, υπάρχουν πλοία τα οποία δεν έχουν πληρώσει την ασφάλειά του κτλ. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για του οποίου μια μικρή ναυτιλιακή εταιρεία, και λέω ότι είναι μικρέ εταιρείε, να μην έρθουν σε επαφή και να μην καταγράψουν τα πλοία μα στη διαδικασία τη Αταλάντα. Αλλά θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να του πείθουμε και σε ό,τι αφορά τι Σεϊχέλε και την Κένια και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πάρα πολύ σαφή ότι έχουμε εξασφαλίσει ότι θα υπάρχει υποστήριξη στι αρχέ των χωρών αυτών σε ό,τι αφορά τους απαραίτητους πόρους, την ύπαρξη συνηγόρων υπεράσπισης για τους πειρατές κτλ. Και όλα αυτά βέβαια θα πρέπει να παρακολουθηθούν και παρακολουθούνται πράγματι από την ομάδα μας. Για όλους αυτούς τους λόγους, αν μπορώ λοιπόν να συνοψίσω, επειδή ξέρω ότι έχετε να αντιμετωπίσετε και άλλα θέματα, δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε σε τρει μήνε. Εντάξει, τέρμα η πειρατεία, το λύσαμε το πρόβλημα αυτό. Θα ξεκολουθεί να ενδυμεί η πειρατεία στην περιοχή αυτή. Οπότε όλοι μας, είτε είναι οι επικεφαλής της ε, ναυτικής δύναμης, είτε είναι οι φορείς της αλληλείας, είτε είναι οι φορείς ναυτιλιακής όλοι από κοινού θα πρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα πού βρίσκονται οι κίνδυνοι, να εξασφαλίσουμε την σωστή διαδρομή που ακολουθούμε να ξέρουμε πού είναι οι περιοχές που είναι πιο ευαίσθητες για να λειτουργήσουμε, να πάρουμε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για να μειώσουμε τον κίνδυνο, είτε σε εθνικό επίπεδο είτε σε αταλαντικό επίπεδο και ελπίζουμε ότι αυτό θα μειώσει και τον αριθμό των πειρατικών ενεργειών. Euh, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίασή σας ε, κύριε Ναύαρχε και γιατί μας απαντήσατε και σε όλες αυτές τις ερωτήσεις, ε, τις πολύ συγκεκριμένε. Ενδεχομένω ο πρόεδρος Σίμψον να ήθελε να πει κάτι πριν φύγετε και ο Αλέν Καντέκ, ε, ε, γιατί συνδιοργανώνουμε την ε, συγκεκριμένη ακρόαση. Σύντομα, κύριε Πρόεδρε, και εγώ να ευχαριστήσω τον υπονάβαρχο λοιπόν για την παρουσίασή του και τις απαντήσεις που έδωσε και να επαναλάβω αυτά τα οποία είπα. Εάν θεωρεί πως μπορούμε να βοηθήσουμε με κάποιον τρόπο, στις επαφές του με το εμπορικό ναυτικό, ευχαρίστω. Εδώ είμαστε. Ειδικά εάν ε, είναι να ενθαρρύνουμε τα εμπορικά πλοία να δηλωθούν σε εσά. Και θα διευκολυνθεί και η δική συμβουλία και αυτή θα είναι πιο ασφαλή. Oui, merci, Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον υπονάβαρχο για τις ε, επεξηγήσεις του. Πραγματικά, κατά τη γνώμη μου, ήταν απαραίτητες. Ήταν ενδιαφέρουσα αυτή η ανταλλαγή απόψε, αλλά και πολύ απαραίτητη. Όσον αφορά τα αλλιευτικά σκάφη, από ό,τι κατάλαβα, ο καλό συντονισμό ε, μεταξύ των διαφόρων μηχανισμών είναι σημαντικό, το είπατε κι εσεί. Κάθε χώρα έχει το μηχανισμό τη ε, και οι Γάλλοι και οι Ισπανοί ειδικότερα, γιατί αυτού αφορά κυρίω το ζήτημα, ότι είναι τεράστιε οι αποστάσει ε, για την επιχείρηση Αταλάντα και είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπερασπιστούμε ολόκληρη την περιοχή. Καταλαβαίνω τις ε, ανησυχίες ε, του συναδέλφου ε, που είπε προηγουμένως μπορούμε να βοηθήσουμε τα σκάφη λόγω, ανάλογα με, την, με το πόσο ευάλωτα είναι να τα θεωρήσουμε κατηγορίας 3. Ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσουμε οπωσδήποτε τον διάλογο με την Επιτροπή σας για αυτή την τυχή. Αυτό το οποίο θα έλεγα, ευχαρίστως η Επιτροπή να έρθει στο στρατηγείο μας, στο Northwood, να δει τι κάνουμε ακριβώς, για να διαπιστώσετε πως καταβάλουμε κάθε προσπάθεια. Και ευχαριστώ να συνεργαστούμε μαζί σας. Ευχαριστώ. Θα έρθουμε τώρα στο επόμενο θέμα που είναι η ρίζα του προβλήματος. Σας περιμένω, σας ζητώ λίγα λεπτά διακοπής ώστε να έρθουν οι άλλοι προσκεκλημένοι μας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Νάβαρχε και καλή επιτυχία στην αποστολή σας.

Αγαπητοί συνάδελφοι, επανερχόμαστε στην ε, συζήτηση. Διευρύνουμε λιγάκι το, την εμβέλεια του θέματος, γιατί ασχολούμαστε γενικότερα με τη Σομαλία. Αναφερθήκαμε στο πρόβλημα της πειρατείας. Αλλά επέκεινα του προβλήματος αυτού υπάρχουν και σημαντικοί λόγοι αστάθειας στη Σομαλία, κάτι το οποίο μας εμπλέκει όλους. Για το θέμα αυτό γνωρίζετε ότι έχουν γίνει και συνεχίζονται να γίνονται συζητήσεις μέσα στους κόλπους του Συμβουλίου για να δούμε αν έχει νόημα να αναπτύξουμε μια ενέργεια της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας προς την υπεράσπιση του, της προσωρινής ομοσπονδιακής κυβέρνηση με τη δημιουργία δυνάμεων ασφαλεία. Αυτό είναι το θέμα το οποίο θα ήθελα λοιπόν να αντιμετωπίσουμε. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Χαρτ Τσέλ, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος τη Σουηδικής Προεδρίας και μετά στον προσωπικό εκπρόσωπο του Χαβιέ Σολάνα, τον κύριο Σουάνα και μετά ο κύριο Μούντα από την Κομισιόν για να μας εξηγήσει λιγάκι πού βρίσκονται τα πράγματα, ποιε είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες πρέπει να προβλεφθούν και σε ποιε συνθήκες. Έχετε το λόγο κύριε Χάρτσελ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω στην υποεπιτροπή σας και συγχαρητήρια και για το επίκαιρο της συζήτησης δεδομένου του ότι οι συζητήσεις ε, των Υπουργών ε, Άμυνας ε, είναι προγραμματισμένες για αύριο. Τώρα, όταν μιλάμε για τη Σομαλία, υπάρχει σαφής σύνδεση με την συζήτηση που μόλις ακούσαμε. Ε, την επιχείρηση Αταλάντα δηλαδή και την καταπολέμηση της πειρατείας. Όπως επιβεβαίωσε και ο Ναύαρχος, εάν μπορούμε να κάνουμε κάτι χρήσιμο για να βοηθήσουμε την σταθερότητα στη Σομαλία, αυτό θα έχει και θετική επίδραση στην αποστολή. Αλλά βεβαίως για το ζήτημα που μας απασχολεί τώρα. Τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Σομαλία. Το ζήτημα είναι ευρύτερο από την πειρατεία. Ξέρετε πως η κατάσταση τους τελευταίους δύο μήνες ε, είναι η εξή. Έχουμε μια μεταβατική ομοσπονδιακή κυβέρνηση με την οποία μπορούμε να συνεργαστούμε και χρειάζεται την υποστήριξή μας για, για να στηριχθεί. Και είχαμε τη διάσκεψη των δωρητών τον περασμένο Απρίλιο, μια σημαντική αφιτηρία. Κατά διάρκεια λοιπόν αυτή τη διάσκεψη ε, και των συζητήσεων που ακολούθησαν, ήταν σαφέ πω η Ευρωπαϊκή Ένωση συλλογικά θεωρούσε πω υπάρχει τώρα μια ανάγκη δράση. Το ίδιο ακούσαμε και από άλλους διεθνεί διεθνείς φορείς. Ε, ξέρετε πως έχουμε την δύναμη της Αφρικανικής Ένωσης επιτόπου, αλλά και από πλευράς ΟΗΕ και είπα υπάρχει ενδιαφέρον να γίνει κάτι. Ε, από κοινού να κάνουμε κάτι. Ένα ενδιαφέρον αυξανόμενο. Το πρώτο βήμα μετά την διάσκεψη των δωρητών του Απριλίου, όταν ξεκινήσαμε σοβαρά να δουλεύουμε, ήταν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του περασμένου Ιουλίου, που ήταν κάπως έτσι μια δήλωση του τι θα ήθελε να επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την πολύπλοκη κατάσταση στη Σομαλία. Τα συμπεράσματα αυτά κατά βάση επαναλάμβαναν πως ε, θέλουμε να κάνουμε κάτι, να συνεργαστούμε με κάποιους άλλους σε αυτή την προσπάθεια και όλα αυτά το στομότερο δυνατόν. Και ξεκαθάριζαν πως ε, ο μόνος τρόπος για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την διεθνή κοινότητα να επιτύχουν τους στόχους τους είναι να γίνει αυτό μέσω μιας συνολικής προσέγγισης. Δηλαδή πρέπει να αντιμετωπίσουμε πολλά ζητήματα τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Τα ακολούθησε μια διερευνητική αποστολή της Προεδρίας, της Γραμματείας του Συμβουλίου, δηλαδή του στρατηγού Ζωανά εδώ πέρα, και της Κομισιόν και είχαμε μια επιτυχία μέχρι στιγμής, το πώς καταφέραμε δηλαδή εμείς οι τρεις να αναλογιστούμε τα πράγματα και να καταλήξουμε σε κάποιες ιδέες. Επίσης αυτή η κοινή διερευνητική αποστολή που ήταν ένα ταξίδι στην περιοχή και μιλήσαμε με όλους ε, τους ε, φορείς εκεί πέρα έγινε πριν λάβει κάποια απόφαση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε ήταν μια αποστολή στην οποία είχαμε μια ανοιχτή συζήτηση από πλευρά Ένωση με όλου του ενδιαφερομένους ανοίξαμε τα χαρτιά μας για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Όπως ε, ξέρετε η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ήδη ενεργή στην Σομαλία. Είμαστε ο μεγαλύτερος δωρητής ε, ανθρωπιστικής βοήθειας. Είμαστε στη Διεθνή Ομάδα Επαφής και συνεργαζόμαστε στενά για να δώσουμε οικονομική στήριξη στην αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης. Και καθώς πλησιάζουμε στα επόμενα βήματα, για να δούμε συγκεκριμένα τον τομέα της ασφάλειας, για το τι μπορεί να γίνει για να δώσουμε καλύτερη, μεγαλύτερη ασφάλεια έχουμε αφενός κατά νου το ότι πρέπει να δράσουμε γρήγορα, αλλά και με σοφροσύνη. Γιατί αν κάνουμε κάποιο λάθος, δεν θα χάσουμε μόνο χρόνο και χρήμα, αλλά διακινδυνεύουμε να γίνει κάτι που θα είναι αντιπαραγωγικό. Τώρα, επειδή έχουμε αύριο το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και το Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας, που θα προγραμματίσει τις ε, αποστολές εκπαίδευσης των Σομαλικών Δυνάμεων Ασφαλείας. Ε, πιθανότατα αύριο θα λάβουμε αυτή την ε, απόφαση για να ε, ενισχύσουμε περαιτέρω το σχεδιασμό μας closely with the partners that και να συνεργαστούμε πιο στενά με τους εταίρους μας για να έχουμε μια επιτυχία αλλά πρέπει να είναι σαφές πως αυτή τη στιγμή η αυριανή απόφαση δεν σημαίνει πως αποφασίζουμε κιόλας πως θα έχουμε μια δράση ΚΕΠΑ. Απλά είναι ένα βήμα ακόμα για να διασφαλίσουμε πως θα έχουμε ευκολότερη πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειαζόμαστε και να ζητήσουμε βεβαίως δεσμεύσεις ε, που θα χρειαστεί για να επιτύχουμε αφενός έχουμε δηλαδή την δέσμευση που θα αναζητήσουμε από την για το ποιος θα είναι ο δικός ο ρόλος στην εκπαίδευση για να λάβουμε για να καταλήξουμε σε μια εκπαίδευση του Ομαλικού στρατού και την ευθύνη τους για το πώς θα οικοδομηθεί μια ευρύτερη δομή ασφαλείας γύρω από την γύρω από τη μεταβατική ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Συνεργαζόμαστε επίσης με την Αφρικανική Ένωση και την δύναμή της εκεί πέρα για να δούμε ποιο ρόλο θα αναλάβει για να μας βοηθήσει στην εκπαίδευση αυτή. Γιατί αυτή είναι επιτόπου. Δεν έχει νόημα να εκπαιδεύουμε σομαλούς στρατιώτες εάν δεν είμαστε σίγουροι πως θα ενταχθούν αυτοί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που θα υποστηρίζει την ε, ομοσπονδιακή μεταβατική κυβέρνηση. Γι' αυτό χρειαζόμαστε την Αφρικανική Ένωση, τη δύναμή της εκεί πέρα να μας βοηθήσει. Ε, Κάποια άλλα ζητήματα για το ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο και τον ρόλο της μεταβατικής κυβέρνησης. Υπάρχει μια μεικτή Επιτροπή Ασφαλείας που λειτουργεί στο Ναϊρόμπι, όπου η διεθνής κοινότητα βρίσκεται σε επαφή, δηλαδή ΟΗΕ, ΗΠΑ Ευρωπαϊκή Ένωση, Αφρικανική Ένωση, θα αποτελέσει λοιπόν έναν κόμβο και θέλουμε εκεί να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με τη μεταβατική κυβέρνηση και πρέπει, όπως σας είπα, να δεσμευτεί και η κυβέρνηση γι' αυτό. Ένα άλλο σημαντικό ορόσημο που θα ακολουθήσει είναι η αξιολόγηση του τομέα ασφαλείας που έγινε υπό την αιγίδα του ΟΗΕ με στήριξη ΕΙΠΑ και λοιπόν που ελπίζουμε ότι θα μας δώσει μια γενική εικόνα για τις, ασφα... για τις ανάγκες του τομέα ασφαλείας και επίσης ε, πιθανές περαιτέρω δράση για το πώς θα γίνει η κατανομή εργασίας μεταξύ των διαφόρων φορέων τη διεθνού κοινότητα και για το τι θα γίνει όσον αφορά την πιθανή εκπαίδευση και πώς θα ενταχθεί σε μια ευρύτερη εικόνα. Θα σταματήσω εδώ. Αυτά από πλευράς Προεδρίας. Έχουμε αναλάβει κάποια σημαντικά βήματα. Δεν έχουν ληφθεί επίσημε αποφάσει. Είναι δύσκολη η κατάσταση, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι να κινηθούμε γρήγορα δεδομένη τη κατάσταση. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ, κύριε Άρτσελ. κύριε Ζωάννα, αν θέλετε να λάβετε το λόγο, να μας διαφωτίσετε κι εσείς για την κατάσταση ασφαλείας και την ευρύτερη περιφερειακή κατάσταση δεν ξέρω αν μπορώ να σας ε, δώσω περισσότερες ε, πληροφορίες γιατί η κατάσταση είναι πάρα πολύ πολύπλοκη. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι να προσπαθήσω να σας διαγράψω το γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εργαζόμαστε. Είτε το θέλουμε, είτε όχι, να συμμετάσχουμε σε αυτή την υπόθεση. Πρέπει να δημιουργηθούν οι δυνάμεις ασφαλείας στην Σομαλία από τον ΝΑΤΟ. Εδώ είναι σαφές ότι θα προχωρήσει αυτό. Και το ερώτημα είναι ποιο είναι το γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούμε. Πρέπει να ξεκινήσουμε από το έργο το οποίο αναφέρθηκε της ομάδας εργασίας για την αξιολόγηση του συστήματος ασφαλείας στη Σομαλία. Η μελέτη αυτή η οποία διεξήχθη από τα Ηνωμένα Έθνη, τους Αμερικανούς και τη διεθνή κοινότητα με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είχε σαν στόχο μαζί με τους Σομαλούς να δούμε πώς λειτουργεί το σύστημα ασφαλείας στη Σομαλία. Ξεκινώντας από τις ένοπλες δυνάμεις, τρόπος του Λέγιν, μέχρι το σύστημα ελέγχου των τελωνίων σοφρονιστικά καταστήματα, αστυνομία, υπουργεία άμυνας, χρηματο, χρηματοδότηση αυτών των ζητημάτων ασφαλείας. Όλα αυτά γίνονται εδώ και δύο μήνες. Τρεις μήνες. Μας λένε ότι στο τέλος Νοεμβρίου θα βγουν τα πορίσματα και τα συμπεράσματα. Ελπίζω θα γίνει αυτό. Και ξεκινώντας από αυτήν την εργασία, η οποία γίνεται για πρώτη φορά με αρκετά ευφύ τρόπο γιατί έχει αντιμετωπίσει το σύστημα ασφαλείας υπό την ευρύτερη δυνατή έποψη. Στη συνέχεια ανέπλεξε από την αρχή τις σομαλικές αρχές, οι οποίες είναι πάντα ενήμερες για την πρόοδο των εργασιών. Εγώ ήμουν παρόν σε συναντήσεις όπου παρουσιάστηκαν τα θέματα αυτά. Υπήρχε ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, ο Υπουργός ε, Εσωτερικής Ασφάλειας, ο Αρχηγός Υπηρεσία ε, Πληροφοριών, διάφοροι, εν πάση περιπτώσει, αξιωματούχοι, οι οποίοι στην πραγματικότητα δεν εκπροσωπούν και πολλά πράγματα, αλλά είναι παρόντες πάντα και επιμελείς. Η διαδικασία πάντως ενσωμάτωσης της ευθύνη της ε, Σομαλίας σε αυτά τα θέματα προχωρεί. Είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε εταίρους οι οποίοι δεν είναι κατά αναγκή θεσμικοί εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών στη Σομαλία και εκπροσώπους της διεθνούς κοινότητος σε αυτή τη διαδικασία. Όταν τελειώσει λοιπόν αυτή η διαδικασία θα έχουμε για πρώτη φορά ένα σχέδιο το οποίο θα μπορέσει να ληφθεί υπόψη πλήρως από τις Σομαλικές αρχές. Δεν υποχρεωμένες βέβαια να δεχτούν αυτές τις προτάσεις, αλλά εφόσον συμμετέχουν στην έκθεση αυτή, πιστεύω ότι θα μπορέσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα να αντιμετωπίσουν αυτή την έκθεση. Και μετά θα πρέπει να λάβουν χώρα μερικές δραστηριότητες, οι οποίες θα έχουν σε στόχο να αντιμετωπίσουμε σε κάθε σχετικό τομέα τις συστάσεις αυτές για να δημιουργήσουμε στρατιωτικές δυνάμεις ασφαλείας, αστυνομικές δυνάμεις, σύστημα δικαστικό, σοφρονιστικό, τελωνιακό, τα πάντα. Μέσα στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει μέσα στα πλαίσια της αποστολής αξιολόγησης και συγχρόνως δείχνουμε ήδη το ενδιαφέρον μας για ορισμένα τμήματα αυτών των συστάσεων που είναι καταρχήν ο στρατός της Σομαλίας αλλά και η αστυνομία στη Σομαλία, το σομαλικό σύστημα δικαιοσύνης κτλ. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει ήδη κάποια πρόοδο στι εργασίε μα. Δεν μιλώ για αυτά που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά σίγουρα έχουμε προχωρήσει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα να εργαζόμαστε για τα θέματα της αστυνομία κτλ. Και μέσα στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να ενσωματώσουμε το τι γίνεται για να αντιμετωπίσουμε τα αίτια της πειρατείας. Γιατί θα πρέπει τα απορίσματα αυτά τα οποία δεν γνωρίζω ακόμα να προτείνουν ένα σύστημα για να προστατεύει τις θάλασσες της Σομαλίας, να υπάρχει ένα λιμενικό σώμα. Επομένως αυτό το γενικό πλαίσιο αρχίζει να διαγράφεται σε ό,τι αφορά τις στρατιωτικές δυνάμεις. Ξεκίνησαν οι προσπάθειες με διμερείς πρωτοβουλίες, με συμμετοχή κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Γαλλία στο Τζιμπουτί και άλλοι, οι οποίοι έχουν εκπαιδεύσει αξιωματικούς και υποξιωματικούς. Έχει ήδη καταρτιστεί ένα τάγμα Σομαλικού στρατού και στην Καμπάλα εκπαιδεύεται το δεύτερο τάγμα. Επίσης και η εκπαίδευση δυνάμεων ασφαλείας περιλαμβάνεται σε αυτό το πλαίσιο. Μου λέτε θα είμαστε συνεπείς με αυτά τα οποία λέει η έκθεση αξιολόγησης. Θα περιγράψει τα θέματα του Σομαλικού στρατού θα πει χρειαζόμαστε μια ταξιαρχία με πυροβολικό τόσο χιλιοστών κτλ. Αυτά που κάνουμε εμείς είναι μονάχα το ένα ελάχιστο, μια ελάχιστη ψηφίδα του, των γενικών αναγκών της Σομαλίας. Επομένως δεν νομίζω θα επηρεάσουμε αυτό το οποίο θα πει η έκθεση. Δεύτερον, να μείνουμε σε ένα καθαρά στρατιωτικό επίπεδο. για νησόμ, η αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης, προσπάθησε να εκπονήσει ένα πρόγραμμα για την εκπαίδευση των δυνάμεων ασφαλείας στη Σομαλία. Η εργασία αυτή είναι στην Αϊρόμπη με συμμετοχή και Βρετανών αξιωματικών και κατέληξαν σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για το οποίο δεν ε, έχουμε να κάνουμε κάποια, ε, αν θέλετε, παρατήρηση να κάνουμε. Γενικά οι συστάσεις αυτές της ΑΝΙΚΟΜ θα ληφθούν υπόψη, αν υπάρχει πράγματι θέληση να γίνει κάτι, μέσα στα πλαίσια των ε, προτάσεων λοιπόν αυτής της ε, έκθεσης της ε, Αφρικανικής Ένωσης, ώστε όλες αυτές οι δράσεις οι οποίες γίνονται, οι εκπαιδευτικές δράσεις που γίνονται σε διμερές επίπεδο, να γίνονται με το ίδιο σχολικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με την ίδια διαδικασία, ώστε να είναι όλα απόλυτα συνεκτικά. Έτσι, χάρη σε όλα αυτά, σας λέω ότι βρισκόμαστε στο σάδιο της μελέτης και αύριο θα γίνει στη συνδιάσκεψη του Καΐρου η, θα ληφθεί η πρώτη απόφαση και από εκεί πέρα μπορούμε να προχωρήσουμε για να δούμε πώς θα φέρουμε σε πέρας όλες αυτές τις ενέργειες. Τώρα για να εξασφαλίσουμε ότι όλα αυτά θα είναι κατανοητά, μαζί με την αποστολή αξιολόγησης έχουμε κάνει το γύρο της περιοχής Συναντήσαμε εκπροσώπους από τη Σομαλία, την Αιθιοπία, την Κένια, πήγαμε και στην Ουγγάντα την προηγούμενη εβδομάδα, ε, και στο Τζιμπουτί φυσικά, στην Αίγυπτο, στην Ασμάρα της Ερυθρέας την προηγούμενη εβδομάδα. Πήγαμε λοιπόν που σας είπα στη Σομαλία και να συζητήσουμε με τους ε, ηθήνοντες. Μιλήσαμε με εκπροσώπους της Αφρικανικής Ένωσης των Ηνωμένων Εθνών, με όλες αυτές τις διεθνείς υπηρεσίες που είναι στην Αϊρόμπη, γιατί όλα γίνονται στην Αϊρόμπη, με τον Αραβικό Σύνδεσμο, προσπαθώντας να έχουμε και την άποψη των χωρών αυτών, γενικά μπορώ να πω ότι όλοι θεωρούν ότι η μεταβατική κυβέρνηση στη Σομαλία μπορεί να μην είναι η βέλτιστη κυβέρνηση που μπορεί να υπάρχει, αλλά τουλάχιστον υπάρχει, δεν υπάρχει εναλλακτική λύση και θα πρέπει να λειτουργήσουμε με αυτά που έχουμε στα χέρια μας. Και εξάλλου όλοι αναγνωρίζουν ότι η Ανισόμ που είναι η αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία είναι ικανοποιητική η δράση θα μπορούσε να κάνει περισσότερο, αλλά δεδομένων των ε, του πλαισίου και του γεγονός ότι κανείς ουσιαστικά δεν θέλει να πάει στη Σομαλία, θα πρέπει να αποδεχτούμε την κατάσταση της ανισόμ. Και όλοι φυσικά συμφωνούν στο να υποστηρίξουμε τις σομαλιακές δυνάμεις ασφαλείας, όχι για να επανελέγξουν το έδαφος που δεν ελέγχουν, γιατί ελέγχουν μονάχα μερικές συνοικίες σε κάποιες πόλεις, αλλά για να δώσει στη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εργαστεί για την ανοικοδόμηση της χώρας αυτής για να μπορούν αυτοί οι οποίοι κάνουν την ανοικοδόμηση να ξέρουν όταν κοιμούνται ότι το άλλο πρωί είναι πιθανό να ξυπνήσουν ζωντανοί. Δεν πρόκειται λοιπόν για τον έλεγχο όλη της χώρας, απλώς να μπορέσει η κυβέρνηση να κάνει το έργο τη χωρί να φοβούνται για τη ζωή του. Επίση, σε σχέση με την επίσκεψη στην Ερυθρέα την προηγούμενη εβδομάδα, ανοίγω μια παρένθεση, είναι η μόνη χώρα που έχει μια σκληρή στάση έναντι της μα μας υπεδέχθη ε, ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, Μίλησα μαζί του για δύο ώρες και τέταρτο. Ήθελε πράγματι να μιλήσει. Γιατί δεν έχει μιλήσει ποτέ με τον πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών που είναι εκεί εδώ και δύο χρόνια. Με εμά μίλησε δυόμιση ώρες, προσπάθησε να μας αγινεύσει, που εμείς δεν ήμασταν τόσο αφελείς για να πέσουμε στην παγίδα, και αναγνώρισε ότι ακόμα και η μεταβατική κυβέρνηση είναι η χειρίστη των κυβερνήσεων με όμικρο γιώτα, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να υπάρξει συμμετοχή στις μελλοντικέ συζητήσεις. Λέει ότι πρέπει να διώξουμε αυτή την κυβέρνηση για να μπορέσουμε να συζητήσουμε με ανθρώπους καλής θέλησης της Σομαλίας στη συνέχεια. Επίσης, επέκρινε τα μάλα την δράση της Ανισόμ, είπε να αλλάξει στάση της Ανισόμ και να μην είναι τόσο μεροληπτική. Βέβαια, όταν έχουμε αυτοκίνητα παγιδευμένα τα οποία κρύγνεται κάθε μέρα, δεν είναι τόσο εύκολο να έχει κανείς μια διαφορετική αντιμετώπιση. Πιστεύω λοιπόν ότι τώρα θα μπορούμε να προβλέψουμε τη δυνατότητα να εργαστούμε. Αν δεν κάνουμε τίποτα λοιπόν, κάποιος άλλος θα το κάνει. η Ουγγάντα είπε ότι θα μείνει στη Σομαλία όσο χρειάζεται και είναι έτοιμη να υποστηρίξει την κατάρτιση των Σομαλιανών δυνάμεων. Ακολουθούν κατά γράμμα το πρόγραμμα το οποίο έχει καταρτήσει η Ανισόμ, λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει καλή επιλογή των υποψηφίων, να είναι καλά εκπαιδευμένοι πρωτού βγουν από το Μογκαντήσιο, να τους ε, συνοδεύουν όταν επιστρέφουν, ώστε να είναι σίγουρο στη Σομαλία ότι θα είναι σε ένα πλαίσιο όπου θα έχουν μια σωστή διοίκηση, ότι θα πληρώνονται και θα υπάρχει κάποιος ο οποίος θα ελέγχει τη συμπεριφορά τους. Δύο εναλλακτικέ επιλογέ υπάρχουν. Είτε του αφήνουν να αναλάβουν εκείνοι τα πράγματα, ε, κάνουμε τα πράγματα όπως ε, γνωρίζουν εκείνοι, βέβαια με την υποστήριξη των Αμερικανών και τη χρηματοοικονομική. Είτε προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την εκπαίδευση επιμένοντας σε ζητήματα τα οποία μας απασχολούν περισσότερα, ε, δηλαδή εκπαίδευση με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνονται πιο σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τώρα, κατά πόσο θα γίνει επιτυχία όλα αυτά, τι να σας πω, δεν ξέρω. Αν η μεταβατική κυβέρνηση έχει το ε, ταλέντο να ανταποκριθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μας χρειάζεται πια, ε, τότε τόσο το καλύτερα. Τόσο το καλύτερο. Μπορεί να μην βελτιωθούν όμως τα πράγματα. Και θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας αυτό. Η ασφάλεια της μεταβατικής κυβέρνησης ε, ε, εξασφαλίζεται από πρώην ε, αρχηγούς. Οπότε πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε γιατί έχουμε ήδη ξεκινήσει. Εμείς είμαστε σε πολύ στενή επαφή με τη μεταβατική κυβέρνηση ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε το γεγονός ότι οι νέε εκπαιδευμένε μονάδες θα έχουν νέες προδιαγραφέ και θα λειτουργούν σε ένα συγκεκριμένο νέο πλαίσιο. ώστε να μην συμμετέχουν οι οπλαρχηγοί που ε, εξακολουθούν ε, να δραστηριοποιούνται ε, αυτή τη στιγμή και βέβαια ελπίζουμε να μην, φύγουμε εμεί και να εξακολουθήσουν να διαστηριοποιούνται οι οπλαρχηγοί γιατί αυτό δεν θα ήταν μια πραγματική επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ και θα ολοκληρώσω εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στρατηγέ, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν και στη συνέχεια θα περάσουμε στη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να εξηγήσω, ε, λέει ο κύριος ε, Ρότζερ Μουρ, πώς ε, συμμετέχουμε εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πειρατεία δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έχει πολύ σοβαρό αντίκτυπο και μάλιστα σε, ένα, σε μια χρονική στιγμή όπου είναι αρκετά ευάλωτες οι χώρες αυτές λόγω της οικονομικής κρίσης ε, την οποία προσπαθούν να αντιμετωπίσουν. Επομένω, η πειρατεία είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα όχι μόνο για την αυτιλία μας αλλά και για την ανάπτυξη των χωρών ε, ε, ολόκληρης της περιοχής αυτής. Η προσέγγιση, όπως ακούσατε, είναι δυτή. Υπάρχει η ανάσχεση και υπάρχει και η εξάλληψη. Η ανάσχεση ε, έχει ως στόχο αυτό που ακούσαμε προηγουμένως. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει την επιχείρηση Αταλάντα ε, με την υποστήριξη των ε, συμφωνιών. Εμείς συμμετείχαμε στις διαπραγματεύσεις και μάλιστα χρηματοδοτούμε εν μέρη τις συμφωνίες με την Γένεια και τις Σεϊχέλες για την κράτηση και την ε, και την δίκη όλων όσων είναι ύποπτοι πειρατείας. Και όσον αφορά τώρα την εξάλληψη, το δεύτερο σκέλος, όπως ε, εξήγησε ο υπονάβαρχος προηγουμένως, ε, πρέπει και στην ξηρά να ε, εργαστούμε. Πρέπει στη Σομαλία να υπάρχει ένα κράτος που λειτουργεί, ένα κράτος δικαίου και για να μπορέσει να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει και σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πρέπει να υπάρχει και δημοκρατία. Και η κατάσταση στη Σομαλία δεν είναι καθόλου έτσι για την ώρα. Επομένως, η δουλειά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Σομαλία ουσιαστικά είναι η οικοδόμηση θεσμών. Είναι κάτι το οποίο η ιδέα του κράτους υπάρχει στο μυαλό του πληθυσμού, αλλά δεν ε, θεωρούν ότι ε, ανήκουν σε ένα κράτος το οποίο λειτουργεί, θεωρούν ότι ανήκουν σε ένα χάος. Οπότε λοιπόν υπάρχουν διάφοροι άξονε επί του οποίου μπορούμε να επικεντρωθούμε για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα κράτο. Ο πρώτο άξονα είναι πολιτικό. Ο δεύτερο είναι η ανάπτυξη, δηλαδή πρέπει. να υπάρχουν κάποιε λογικέ προσδοκίε ε, όσον αφορά το επίπεδο διαβίωση. Το θέμα τη ασφάλεια επίση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και υπάρχει θέμα και της περιφερειακής διάστασης βέβαια, γιατί γνωρίζουμε ότι η Σομαλία βρίσκεται σε μια περιοχή η οποία είναι αρκετά επιρροή, επιρρεπής ε, στις συγκρούσεις, ε, ανήκει στο κέρα τη Αφρική, γνωρίζουμε πολύ καλά ε, πώς είναι η κατάσταση, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου το ανέφερε. Ένας από τους λόγους, ένας από του τρόπους ήταν να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πώς η κάθε χώρα ε, αντιλαμβάνεται την κατάσταση. Προσπαθήσαμε λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο να ε, αποτελούν μέλη της, με, μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος. Όσον αφορά τώρα τη δουλειά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την κατεύθυνση αυτή, Όσον αφορά την ανάπτυξη, που βέβαια είναι ο παραδοσιακός ε, τομέας ε, στον οποίο εργαζόμαστε, 300 εκατομμύρια ευρώ περίπου ε, σε επιχειρήσεις στην Σομαλία αυτή τη στιγμή, το ίμιση 150 εκατομμύρια περίπου αφορά την ανάπτυξη, χρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και 11 εκατομμύρια αναπτυξικών επιχειρήσεων από το μέσο σταθερότητας και Έχουμε επίσης και την υποστήριξη της Αμισόμ, προστασία δηλαδή στις κυβερνήσεις, 95 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή αποκινούμε την Αμισόμ και όσον αφορά τα ανθρωπιστικά 44 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Είναι χαμηλότερο το ποσό, είναι μικρότερο το ποσό, αλλά ούτως ή άλλως η προθεσμία που έχουμε είναι πολύ μικρότερη. Έχει ε, ήδη διατεθεί το ποσό. Τώρα, τι κάνουμε όσον αφορά την ανάπτυξη Προσπαθούμε να επιτύχουμε τη διακυβέρνηση, την εκπαίδευση, την οικονομική ανάπτυξη, ανάπτυξη της υπαίθρου. Και όσον αφορά τη διακυβέρνηση, υπάρχει πάντοτε το πρόγραμμα κράτους δικαίου, το οποίο ε, έχει πρικοδοτηθεί με 13 εκατομμύρια ευρώ. Το ανέφερε και ο στρατηγός Ζωανά. Ε, εργαζόμαστε από κοινού με την ε, για το δικαστικό πρόγραμμα και το αστυνομικό ε, πρόγραμμα ε, και είμαστε κάπως επιτυχείς σε αυτό το τομέα. 29 προγράμματα, 66 εκατομμυρίων ευρώ, 68 εκατομμυρίων ευρώ, σε τρεις περιοχές της Σομαλίας, ε, Σομαλιλάνδη, και Σομαλία και την κεντρική ε, κεντρική δυτική πλευρά, δηλαδή την περιοχή γύρω από το Μογκαντήσου, 46 εκατομμύρια ευρώ ε, τα οποία έχουμε αποσύρει από την ε, κεντρική και νότια Σομαλία γιατί υπήρξαν ε, κάποια λυπηρά περιστατικά. Αποφασίσαμε ότι δεν είναι αρκετά ασφαλές να δραστηριοποιηθούμε στην περιοχή αυτή. Και όσον αφορά τώρα την οικονομική ανάπτυξη και την ανάπτυξη της υπαίθρου, έχουμε 19 προγράμματα στο σύνολο, 42 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό που θα έπρεπε να πω επίσης είναι Αναρωτιέστε πώς γίνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαχειρίζεται προγράμματα σε περιοχές όπου η κυβέρνηση δεν μπορεί να το κάνει. Είναι μία από τις σοβαρές δυσκολίες που έχουμε κατά την οικοδόμηση των θεσμών, γιατί αυτό που χρειαζόμαστε είναι βέβαια να ασφαλίσει η κυβέρνηση να μπορεί να παρέχει υπηρεσίες και δεν είναι βέβαια τόσο παραγωγικά τα πράγματα όσον αφορά ε, την ε, ανάπτυξη θεσμών, ε, όπως θα ήταν αν υπήρχαν μη κυβερνητικέ οργανώσεις, για παράδειγμα. Η κυβέρνηση δεν είναι παρούσα σε μεγάλο τμήμα της κεντρικής και νότιας Σομαλίας ε, γιατί η, Αμισού, η Αμισόμ ανέλαβε δράση επειδή υπήρχε ένα κενό εξουσίας ε, και ένα τμήμα της πολιτικής μας προσέγγισης είναι να τους ενθαρρύνουμε να προσπαθήσουν ε, να ασχοληθούν με όλους αυτούς τους τομείς, κάτι το οποίο δεν θα ήταν μάλλον, δεν θα πρέπει να είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και βέβαια Θα ήθελα να μιλήσω και λίγο για τα κράτη-μέλη, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτως ή άλλως έχει κάποια προγράμματα για τη Σομαλία. Έξι κράτη-μέλη μας υποστήριξαν και η Νορβηγία. Είχαμε ένα κοινό προγραμματισμό. Οπότε τώρα τα συνολικά ποσά είναι περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ κατέτος για τη Σομαλία 150, τα μισά δηλαδή, προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 85 εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και νομίζω ότι θα σταματήσω εδώ για να δώσω περισσότερο χρόνο σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ. Πρωτού δώσω το λόγο στους συναδέλφους οι οποίοι θέλουν να ζητήσουν τον ίδιο αυτό το λόγο, θα ήθελα και εγώ να αναφερθώ σε ένα ερώτημα σε ό,τι αφορά τη Σομαλιλάνδη και την περιοχή του Πούντ. Γιατί μέσα στο συνολικό χάος υπάρχουν περιφερειακές οντότητες οι οποίοι φαίνονται λειτουργικότερες των άλλων, πιο σταθερές, πιο... πιο ισχυρές από τις άλλες. Είναι γεγονός ότι η προσωρινή κυβέρνηση θα σεβαστεί το καθεστώς αυτών των περιοχών, των περιφερειακών αυτών οντοτήτων. Όταν μιλάτε για προγράμματα λοιπόν εκπαίδευσης για την, στο έδαφος της Σομαλίας, θα μπορέσει και η, η κεντρική κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει αυτές τις περιοχές. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά την Ερυθρέα. Αναφερθήκατε σε αυτή τη συνάντηση με τον ηγέτη της Ερυθρέας. Από πολλές απόψεις η Ερυθρέα από τις άλλες χώρες της περιοχής την αντιμετωπίζανε σαν να είναι ο άτακτος κατά κάποιο τρόπο της γειτονιάς και όχι ένα σταθεροποιητικό στοιχείο για τη Σομαλία. Αναφερθήκατε στο θέμα αυτό με τρόπο αρκετά επιφυλακτικό βέβαια. Θεωρείτε ότι αυτό είναι συγκυριακό ή είναι απλώς μια μακροχρόνια γραμμή που θα ακολουθηθεί από την Ερυθρέα. Και θα ήθελα επίσης να ξέρω ποια είναι τα προγράμματα τα οποία εφαρμόζει η Κομισιόν στην Ερυθρέα σχετικά. Θα δώσω πρώτα το λόγο στην κυρία Μπραντ Νέαρ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχω δύο ερωτήματα και πρέπει να είμαι σαφής. Η παρουσίαση η οποία έγινε δεν με έπεισε ιδιαίτερα ότι έχει μεγάλο νόημα να υποστηρίξουμε μια νέα αποστολή στην περιοχή αυτή. Δεν είμαι σίγουρος ότι η προσθέμενη αξία της ευρωπαϊκής αυτής αποστολής θα είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Δεν ξέρω αν έχει νόημα να γίνει αυτή η αποστολή. Το επιχείρημα ότι αν δεν το κάνουμε εμείς θα το κάνουν οι άλλοι εγώ δεν ε, πείθομαι από αυτό το επιχείρημα σε σχέση με την εκπαίδευση των δυνάμεων στη Σομαλία και θέτω αυτό το ερώτημα γιατί από ό,τι καταλαβαίνω βλέπω ότι η Κομισιόν κάνει πάρα πολλά για την ανάπτυξη της αστυνομίας αλλά όταν μιλάμε για δυνάμεις ασφαλείας μιλάμε και για τον στρατό. Και τίθεται το θέμα της εκπαίδευσης του στρατιωτικού, των στρατιωτικών δυνάμεων. και θα ήθελα να ξέρω αυτοί οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν στις ε, ενέργειες κατάρτισης που αναφέρατε ήταν αστυνομικοί ή περισσότερο στρατιωτικοί. Τίθεται επίση το ερώτημα του πώς θέλετε να εξασφαλίσετε ότι τα άτομα αυτά μετά θα πληρώνονται, θα είναι ενσωματωμένα στο σύστημα. Εγώ δεν μπορώ να κατανοήσω πολύ καλά τι έχει προβλεφθεί να γίνει σε αυτήν την περίπτωση. Ίσως μπορείτε να μου πείτε κάτι περισσότερο για το θέμα αυτό, το οποίο για μένα είναι κομβικό για την επιτυχία αυτής της αποστολής. Τέλος, ξέρουμε ότι δεν έχουμε ακόμα τα πρόσθετα άτομα τα οποία έχει ζητήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το Αφγανιστάν, για εκπαίδευση εκεί και τώρα έχουμε μία νέα αποστολή την οποία θέτουμε σε κίνηση χωρίς να έχουμε καλύψει τις προηγούμενες προτεραιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήταν η, το Αφγανιστάν. Δεν ξέρω λοιπόν αν είναι δικαιολογημένο να ανοίγουμε νέα μέτωπα όταν δεν έχουμε κλείσει τα παλιά. Δεν βρίσκω λοιπόν πολύ ικανοποιητική την εξήγηση που μου δίνεται. Ευχαριστώ. Άλλα ερωτήματα, ο κ. Γκουαλτιέρη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να πω ότι αυτά που ακούσαμε προφανώς γεννούν κάποια ερωτηματικά και θα ήθελα και εγώ να έχω περισσότερες λεπτομέρειες, περισσότερες διευκρινήσεις. Δεν χωρεί αμφιβολία και το είδαμε πολύ καλά και στην προηγούμενη συζήτηση που κάναμε με τον ε, υπονάβαρχο Χάντσον ότι είναι απαραίτητο να μην, να μην περιορίζουμε τη δράση μας σε μια αντιμετώπιση στη θάλασσα των πειρατών, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις ρίζες του φαινομένου αυτού και να ενισχύσουμε τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ίδια τη Σομαλία. Συγχρόνως είναι αναμφίβολο ότι η κατάσταση επιτόπια είναι τέτοιου είδους που τα προβλήματα της ασφάλειας είναι, αν θέλετε, η επίλυση των προβλημάτων, δηλαδή ασφάλειας, είναι προαπαιτούμενα για τη δημιουργία μιας κυβέρνησης, ενός κράτους κτλ. Αλλά συγχρόνως δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε ότι το γεγονός είναι ότι είναι πολύ περιορισμένη εντολή αυτής της δυνητικής εντολής, γιατί δεν νομίζω ότι είμαστε στο επίπεδο της εκκίνησης αυτής της αποστολής, κάνουν πολύ δύσκολο να καταλάβουμε σε ποιο βαθμό αυτή η αποστολή μπορεί να είναι σε θέση να επηρεάσει μια διαδικασία η οποία, όπως αναφέρεται, ουσιαστικά γίνεται αφεαυτής χωρίς την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να καταλάβω λοιπόν καλύτερα μέσα στα πλαίσια αυτών των προγραμμάτων που αναφέρεται Ποια είναι η σχέση μεταξύ αυτών των διμερών ενεργειών που γίνονται από τις ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι σχέση έχουν με την πραγματική ανάγκη που υπάρχει για την εκπαίδευση δυνάμεων ασφαλείας προς το όφελος της προσωρινής κυβέρνησης. Επομένως, το ερώτημα μου είναι πώς αυτή η αποστολή μπορεί δυνητικά να επηρεάσει την εκπαίδευση αυτών των δυνάμεων ασφαλείας στη Σομαλία. Και σε ποιο βαθμό αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα στα πλαίσια μιας γενικότερης πολιτικής αξιολόγησης για τη δυνατότητα να επιτευχθεί εσωτερική ισορροπία στο κράτος της Σομαλίας, να υπάρξει ισορροπία μεταξύ κρατική οντότητα και περιφερειακής ισορροπία και εγγραφή σε ένα ευρύτερο περιφερειακό πλαίσιο. Ευχαριστώ. Μπουτικόφερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θέλω να κάνω κάποιες έτσι ερωτήσεις με κάποιο σκεπτικισμό δεν κατάλαβα ακριβώς τι θα αποφασίσουν αύριο οι Υπουργοί Εξωτερικών. Θα αποφασίσουν κάτι ή θέλουν να προετοιμάσουν μια απόφαση ή θέλουν να συζητήσουν την προετοιμασία μιας απόφασης. Τι είναι η συζήτηση αύριο, τι θα γίνει ακριβώς. Δεύτερον, εγώ κατάλαβα στο επίπεδο των μέσων πως πρέπει να εκπαιδευτούν δυνάμεις ασφαλείας δεν κατάλαβα ποιος είναι ο πολιτικός στόχος. Ποιο χρονικό ορίζοντα έχει αυτός ο πολιτικός στόχος και όταν εμπλακούμε πώς θα φύγουμε από εκεί. Και δεν κατάλαβα γιατί πέρα από αυτά τα οποία κάνει η Γαλλική Δημοκρατία για την εκπαίδευση των δυνάμεων ασφαλείας, γιατί τώρα πρέπει να εμπλακεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση επιπλέον. Γιατί δεν λέμε. Ε, πρώτα απ' όλα ας εφαρμόσει αυτά που θέλει η Γαλλική Δημοκρατία και έχει μετά άλλε προτεραιότητες η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν κατάλαβα. Ποιες προσδοκίες σταθεροποίησης έχετε όταν στηρίζετε αυτή τη μεταβατική κυβέρνηση. Ο κύριος Ζωανά είπε σχεδόν επιλέξει πως εάν ρωτούσαμε τη μεταβατική κυβέρνηση θα μας λέγανε δεν σας χρειαζόμαστε. Ε, είναι έξυπνη πολιτική αυτή. Δηλαδή εμείς να πιέσουμε και να έχουμε αυτό ως βάση στρατιωτικής εμπλοκής. Αυτά. Ερωτήσεις επί ερωτήσεων. Okay, um, start out trying to... Θα ξεκινήσω εγώ προσπαθώντας να απαντήσω τις ερωτήσεις όσο μπορώ και μετά και ο Ρότζερ και ο στρατηγός Ζωανά θα απαντήσουν. Για την πρώτη ερώτηση, τον ρόλο της περιοχής του Πούντ και της Σομαλιλάνδης. Είναι σαφές, ε, ερχόμαστε στο συνολικό ερώτημα του τι πρέπει να γίνει στη Σομαλία για να έχουμε επιτυχία. Και αυτό είναι να εξασφαλίσουμε πως η εκπαίδευση πρέπει να ενταχθεί σε ένα γενικότερο πλαίσιο και όταν έχουμε δεσμεύσεις από τη μεταβατική ομοσπονδιακή κυβέρνηση όσον αφορά τον ρόλο της στην εκπαίδευση, στην ασφάλεια, πρέπει να συνεργαστούμε μαζί τους για να συνεχίσουν στην διαδικασία πολιτικής συμφιλίωσης και βεβαίω εκεί υπάρχουν διαφορετικές διαστάσεις. Υπάρχει κατάσταση στο Νότο αλλά και η κατάσταση στην περιοχή του Πούντ και της Ομαλιλάνδη και κοιτάμε τώρα το τι μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με την εκπαίδευση και το πού πρέπει να γίνει εκπαίδευση και δεν κοιτάμε να γίνει αυτό εντός ε, της Σομαλιλάνδης ή της περιοχής του Πούντ αυτή τη στιγμή για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων ασφαλείας μάλιστα, πρέπει να γίνει αυτό αλλού. Και δεν αποκλείεται αυτό το οποίο κάνουμε για την οικοδόμηση του τομέα αυτού στην Σομαλία να γίνει σε ένα ευρύτερο πλαίσιο όταν έρθει η ώρα. the value added of... Τώρα, για το τι προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην εκπαίδευση αναφέρθηκε το τι μπορεί να προσθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ναι, σωστό είναι αυτό, δεν πρέπει να το υποτιμάμε. Είναι πολύ σημαντικό οι πτυχές αυτές να αποτελέσουν τμήμα της οποιασδήποτε εκπαίδευση με τους ε, νεαρούς αυτούς σομαλούς. Να εκπαιδευτούν δηλαδή κατά τρόπον ώστε να μην ε, μάθουν μόνο να λύνουν και να δένουν τα όπλα τους, αλλά να αναλάβουν και τις ευθύνες του συζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης, αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η εκπαίδευση αυτή να μπει σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο. Εάν ξεκινήσουμε με την εκπαίδευση, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να συστήσουμε μια συνεργασία με όλους τους εταίρους, όχι μόνο την Αφρικανική Ένωση. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Πρώτα απ' όλα υπάρχει σταθερή συνεργασία με την Αφρικανική Ένωση. Δεύτερον, υποστηρίζουμε αυτή τη στιγμή την Αμισόμ. Και με βάση αυτά υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθεί μια ολόκληρη αλυσίδα είτε από πλευράς ελέγχου προσώπων στη Σομαλία μέχρι την ίδια την εκπαίδευση που, στην οποία θα δοθεί μετά η κατάλληλη συνέχεια. Επιπλέον η εκπαίδευση πρέπει να ενταχθεί στο ευρύτερο πλαίσιο του τομέα της ασφαλείας. The work that's been done. Ο Δε Ρότζερ Μουρ ανέφερε το τι θα γίνει γενικότερα σε σχέση με τη μεταβατική κυβέρνηση την οικοδόμηση δηλαδή ενός κράτους και η οικοδόμηση του κράτους θα αποτελέσει ένα σημαντικό κομμάτι όταν μιλάμε για δομές ασφαλείας. Πρέπει να σκεφτούμε το πώς θα είναι οι δομές αυτές στον τομέα αυτών. Πρέπει να βοηθήσουμε και την κυβέρνηση με κάποιον τρόπο και αυτό χρειάζεται πηγόντως έτσι ώστε η εκπαίδευση αυτή στο τέλος θα έχει κάποιο νόημα ότι θα αποτελέσει δηλαδή ένα μέσο σταθερότητας και θα είναι στη σωστή πλευρά και όχι στη λάθος. Επίσης αναφέρθηκε το ζήτημα των πληρωμών. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε εξετάζουμε διάφορες ε, επιλογές και είπα αυτή τη στιγμή καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες ώστε να βρεθεί ένας μηχανισμός στον Ναϊρόμπι μέσω της PricewaterhouseCoopers ε, που θα λειτουργεί έτσι ώστε πρώτα απ' όλα να υπάρχει λογοδοσία για τα χρήματα και μετά οποιασδήποτε πληρωμές μέσω αυτού του μηχανισμού να φτάσουν στον τελικό αποδέκτη. Και αυτό εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να το δούμε και να δώσουμε συνέχεια. Excellent opportunity to do so, uh, uh, the broad contacts um, and the, the, the, role we are. Και ο ρόλος βεβαίως ο οποίος uh, παίζουμε στην Σομαλία και στην περιοχή πρέπει να οδηγήσει στην συνεργασία, όπως σας είπαμε, τη μεταβατική κυβέρνηση για να γίνουν όλα αυτά. As regards the decision uh, that ministers might be taking to... Οποιαδήποτε απόφαση δύναται ληφθεί υπό τον Υπουργό Εξωτερικών θα πρέπει να εστιάζεται σε μια εθνική ενατένιση του μέλλοντος της Σομαλίας. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα πρώτο εποφελές βήμα ώστε να ξεκινήσει μια νέα διαδικασία σχεδιασμού μέσα στα πλαίσια της ΚΕΠΑ. Όπως είπα όμως αυτό δεν σημαίνει ότι μια απόφαση έχει ήδη ληφθεί για να ξεκινήσει μια τέτοια αποστολή στη Σομαλία. Αντίθετα, αυτό το οποίο επιζητούμε είναι να εξασφαλίσουμε ότι μπορούμε να σχεδιάσουμε μια τέτοια αποστολή με αποτελεσματικό τρόπο, εάν αυτό είναι απαραίτητο. Τέλος, πού θα βάλουμε τους πόρους μας και πώς θα εκπαιδεύσουμε το προσωπικό αυτό στο Αφγανιστάν. Κάτι το οποίο ενδιαφέρει ιδιαίτερα και το δικό μου Υπουργό και πολλούς άλλους Υπουργούς ο Καλμπιλτ μαζί με τον Χαβιέ Σολάνα έχουν κάνει μια μεγάλη προσπάθεια για να αναπτύξουν την EU pol στο Αφγανιστάν. Ο στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι μπορούμε να εκπαιδεύσουμε σωστά τις αστυνομικές αρχές του Αφγανιστάν και χρειάζεται λοιπόν ενίσχυση της EU-POL. Και το ίδιο ισχύει για πάρα πολλές από τις αποστολές μας. Όλες οι αποστολές μας έχουν έλλειψη προσωπικού. Αλλά τίθεται και το ερώτημα του κατά πόσο θα πρέπει να αφήσουμε τους πόρους να χαλιναγωγήσουν τις πολιτικές μας φιλοδοξίες. Και επίσης τίθεται ένα ακόμα θέμα, όταν πρόκειται για το προσωπικό, το οποίο ψάχνουμε να βρούμε για την U-Pol στο Αφγανιστάν. Οι περισσότεροι από αυτούς θα είναι αστυνομικοί ενώ αν μιλάμε για την εκπαίδευση που θέλουμε να κάνουμε στη Σομαλία, έχουμε άλλου είδους κατηγορίες ανθρώπων οι οποίοι θα είναι χρήσιμοι. Επομένως δεν είναι εναλλάξιμοι αυτοί οι πόροι και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο ίδιο πλαίσιο. Ούτως λοιπόν μπορώ να αφήσω το λόγο στον στρατηγό Ζουάνα. Στρατηγέ μου, Απλώς θέλω να σας πω ότι δεν κάνουμε μια επιχείρηση ΚΕΠΑ για να κάνουμε μια επιχείρηση ΚΕΠΑ, για να κάνουμε το κέφι μας ούτως πίν. Υπάρχουν αποφάσεις ηλιμένες οι οποίες μας οδηγούν να μελετήσουμε σοβαρά το τι θέλουμε να κάνουμε για να υποστηρίξουμε και την κυβέρνηση. Ο στόχος μας λοιπόν είναι να εγγραφούμε με απόλυτη σαφήνεια στο πλαίσιο το οποίο υπάρχει σε διεθνές επίπεδο, καταρχήν κάτω από την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και επίσης θα πρέπει να βρεθούμε πίσω από την Αφρικανική Ένωση και στα πλαίσια της εταιρικής σχέσης που έχουμε για τα θέματα ασφάλειας με την Αφρικανική Ένωση. Προτού λοιπόν σκεφτούμε να φτιάξουμε μεταξύ μας μια μικρή ευρωπαϊκή αποστολή, ο στόχος μας ήταν να συνεργαστούμε στενά με την Αμισόμ, με τους φίλους μας στη Σομαλία, με την Αφρικανική Ένωση, ώστε να μην υπάρχει λοιπόν καμία ε, διαφορά απόψεων σε σχέση με τη διαδικασία εκπαίδευσης που στοχεύουμε να κάνουμε. Στη συνέχεια, μέσα σε αυτή την εταιρική σχέση θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια βελτιστοποίηση των χρηματοοικονομικών πόρων που δίνονται στην Αφρικανική Ένωση, παραδείγματος χάρη διευκολύνσεις πληρωμών και να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους πόρους ώστε να τους κατευθύνουμε προς την κατεύθυνση της υποστήριξης της Αφρικανικής Ένωσης για την αποκατάσταση μιας κατάστασης όσο το δυνατόν πιο φυσιολογικής στην Σομαλία. Είναι λοιπόν ένα έργο το οποίο θα βρίσκεται σε στενή σύνδεση με την Αφρικανική Ένωση. Τέτοιου είδους αποστολές δεν φύγουν ήδη οι φυστάμενες διμερείς πρωτοβουλίες. Ο στόχος μας αντίθετα είναι να υποστηρίξουμε όλες αυτές τις διμερείς πολυμερείς πρωτοβουλίες και να τις κατευθύνουμε στην ίδια γραμμή δράσης, να έχουμε κοινούς στόχους, να εργαστούμε μέσα στα πλαίσια των συστάσεων που θα προέλθουν από την αποστολή αξιολόγησης, να υποστηρίξουμε τις αρχές της Σομαλίας, ώστε κάθε μικρό πετραδάκι να μπορέσει να βοηθήσει να χτίσουμε τον κοινό ουρανοξύστη. Έχουμε λοιπόν τη Γαλλική Πρωτοβουλία στο Τζιμπουτί, η οποία ήταν κατά κάποιο τρόπο μια πειραματικού χαρακτήρα αποστολή. Οι ίδιοι οι Γάλλοι και η Ευρώπη φυσικά ίντλησαν τα απαραίτητα συμπεράσματα για το τι θα πρέπει να γίνει στην τροποποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος και επίσης <clears throat> θα πρέπει να πάρουμε τις δύο ελίπουσες ψηφίδες που έχουν να κάνουν με τη στενή συνεργασία με τους Σομαλούς και να μπορέσουμε να δούμε πώς θα προβλέψουμε τη συνέχεια της εκπαίδευσης αυτών των στρατιωτών όταν γυρίσουν στη Σομαλία. Διότι θα δεν έχει νόημα να βάλουμε 800 φαντάρους σε ένα στρατόνα όπου δεν θα τους δίδεται καν μια πληρωμή. Αυτό είναι κάτι το οποίο λοιπόν είναι απαραίτητο να το σκεφτούμε όταν θέλουμε να δώσουμε μια συζήτηση. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε ένας Ευρωπαίος στη Σομαλία. Κανένας μη κυβερνητικό οργανισμός στην Σομαλία παρά μόνο πιλωτικά. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται επιτοπίως και με τους οποίους μπορούμε να έχουμε μια σχέση εμπιστοσύνης είναι η εταίροι μας από την Αφρικανική Ένωση. Αυτοί λοιπόν θα πρέπει να κάνουν την επιλογή, τον θετικό έλεγχο, την, τον ιατρικό έλεγχο, τον αποκλεισμό των ανηλίκων. Όλα αυτά είναι πολύ δύσκολα να γίνουν. Όλα αυτά πρέπει να βασιστούμε στην Αφρικανική Ένωση να τα κάνει και όλα αυτά πάντα σε στενή συνεργασία με τις αρχές της Σομαλίας. Δεν θέλουμε να τους επιβάλλουμε μία λύση. Όχι. Έχουμε συζητήσει με τον Πρωθυπουργό και τους διάφορους υπουργούς για τον καλύτερο τρόπο να επιχειρήσουμε. Αυτοί προφε... προτιμούν να υπάρξει επιτόπια εκπαίδευση. Θεμητό είναι αυτό. Κατανοούν ότι οι συνθήκες ασφαλείας προς το παρόν δεν είναι <clears throat> οι καλύτερες και προς το παρόν θα είναι καλύτερο φαίνεται σε εμά να του εκπαιδεύσουμε αλλού και να του φέρουμε μετά στην, Σουμαρία, στην Σομαλία και για περιοχέ όπω το Πούντλαντ, η υπερχή του Πούντ, είπε ο Πρωθυπουργό ότι θα μπορούσε αυτό το πράγμα να γίνει εκεί. Όλα αυτά λοιπόν δεν στρέφονται κατά τη Σομαλιανή κυβέρνηση. Απλώ θέλω να υπογραμμίσω ότι ο ρυθμό κατάρτισης εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η ανάμειξη των παλαιοσυρών με τους νεοσύλλεκτους, ώστε να μην υπάρξει μια ένταση μεταξύ τους στα πλαίσια των στρατιωτικών δυνάμεων. Και υπάρχουν πολλοί στρατιωτικοί μηχανισμοί, μηχανισμοί πληρωμών οι οποίοι είναι υπό εξέταση. Έχουμε την εμπειρία των ε, Κινέζων και των Αμερικανών και φυσικά της έγκριτης εταιρείας Pricewaterhouse αλλά και Cooper Μπορούμε λοιπόν με τον τρόπο αυτό να προχωρήσουμε προς ε, μια λύση. Καταρχήν πρέπει να βρούμε τα χρήματα, γιατί προς το παρόν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί αυτή και μόνη να χρηματοδοτήσει τη, τους μισθούς των στρατιωτικών. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε κάποια διμερή συμφωνία και υπάρχουν άλλοι εταίροι οι οποίοι μπορούν να πληρώσουν οι Αμερικανοί, οι Λίβοι. Εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι πρέπει να δίνουμε ένα εκατομμύριο δολάρια το μήνα για να μισθοδοτούμε το στρατό της Σομαλίας. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι αυτός ο οποίος θα δίνει τα λεφτά να πιάνουν τόπο τα χρήματά του και φυσικά θα έχει κάθε δικαίωμα να ζητήσει να μάθει πώς χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα χρήματα. Άλλο θέμα είναι να ξέρουμε ότι τα λεφτά αυτά θα φτάσουν στους στρατιώτες. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί εμείς δεν μπορούμε να ελέγχουμε στη θέση της Σομαλίνης κυβέρνησης, δεν μπορούμε να είμαστε επιτοπίως. Θα πρέπει καταρχήν να σεβαστούμε την κυριαρχική ε, εξουσία της Σομαλιανής κυβέρνησης. Γι' αυτό έχουμε επιλέξει αυτόν τον τόσο διάφανο μηχανισμό, τον πιο διάφανο που μπορούμε να έχουμε. Και εξάλλου οι Σομαλοί όλοι λέγονται Ιουσούφ, Αμπτουλά ή κάτι τέτοιο. Δύο-τρία ονόματα έχουν όλοι και τα μοιράζονται μεταξύ του. Δεν μπορούμε λοιπόν να αποφύγουμε τα σφάλματα. Γιατί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση Γιατί λοιπόν δεν αφήνει τη Γαλλία να κάνει κάτι εκεί. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να έχουμε κάποια πρόοδο εκτός αν όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση εμπλακεί στο θέμα αυτό. Είτε συνεχίσουν είτε δεν συνεχίσουν οι Γάλλοι. Εν πάση περιπτώσει και ίσως όχι στις τρέχουσες συνθήκες, σας είπα ότι θέλει να εμπλακεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί θέλουμε να υποστηρίξουμε μια αποστολή, η οποία ήδη ίδια αυτή υποστηρίζει τη μεταβατική ε, κυβέρνηση στη Σομαλία. Και εξαρτώμεθα πάντα από τις αρχές της περιοχής αυτής. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους πόρους και την δυνατότητα χρησιμοποίησή τους στο Αφγανιστάν, εγώ δεν έχω να σας δώσω μία απάντηση. Σαν στρατιωτικός δεν νομίζω ότι μας λείπουν οι πόροι στους ευρωπαϊκούς στρατούς. Είναι απλώς η απόφαση των ευρωπαϊκών στρατών να χρησιμοποιήσουν ένα μέρος των δυνάμεων τους για να τους εμπλέξουν σε μία διαδικασία. Και αν δεν υπάρχουν αρκετά κράτη-μέλη τα οποία θα δώσουν τις δυνάμεις αυτές, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Εγώ πήγα τρεις φορές στο Κονγκό για να δω πώς θα υπάρξει μεταρρύθμιση της κατάστασης εκεί για την ε, βελτίωση της κατάστασης. Μας είχαν υποσχεθεί χίλιους αξιωματικούς, εγώ είδα 40 εκεί λοιπόν, αλλά έτσι γίνεται πάντα. Αυτά πρέπει να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Ευχαριστώ στρατηγέ μου. Κύριε Διευθυντά. Να σχολιάσω δύο πράγματα. Καταρχά υπήρχε μια συγκεκριμένη ερώτηση για την Ερυθρέα είναι λίγο διαφορετικό το θέμα της Ερυθρέας, όπως είπα και προηγουμένως, επειδή υπάρχουν κάποιες περιφερειακές διασυνδέσεις και είναι πολύ σημαντικό να συνδεθούν τα δύο ζητήματα. Η πολιτική μας για την Ερυθρέα είναι κάτι η οποία δεν, είχε, δεν έχει βραχυπρόθεσμα, αλλά μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Παρόλα αυτά, η πολιτική μας ε, έχει να κάνει με το εξή. Η Ερυθρέα στην τελευταία μα επίσκεψη μα είπε ότι θα ήθελε να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια πολιτική για τη Σομαλία και αν υπάρχει βεβαίω θέληση. Είναι προ συμφέρον μας ε, να ε, επενδύσουμε και οικονομικά και από άποψη θέληση. Όσον αφορά τώρα την αναπτυξιακή μας συνεργασία, αυτή τη στιγμή 130 εκατομμύρια έχουμε προβλέψει για ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα 6 ετών από το Ευρωπαϊκό, πρόγραμμα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, 2 δισεκατομμύρια για το κέρας της Αφρικής και η Ερυθρέα δεν θα λάβει πάρα πολύ χρηματοδότηση γιατί ουσιαστικά είναι, ε, είναι γιατί θεωρούμε ότι είναι καλύτερα να είμαστε πιο μετριοπαθείς στις προσδοκίες μας. Ε, τα αποτελέσματα της συνεργασίας μας με την Ερυθρέα είχαν ως αποτέλεσμα 10 με 20 εκατομμύρια ευρώ κατέτος και κυρίως αφορά επισητιστική ασφάλεια που είναι και η βασική ανησυχία της κυβέρνησης. Έχουμε και ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης. Ε, η επισητιστική ασφάλεια θα αφορά και την, και την παραγωγή αλλά και ε, την ε, μεταφορά προμηθειών. Και τώρα θα ήθελα να αναφερθώ στο πολιτικό στόχο της εκπαίδευσης ε, ε, ασφάλειας, δυνάμεων ασφαλείας. Αν θέλουμε να βελτιώσουμε τα πράγματα με την πειρατεία, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με την οικοδόμηση θεσμών, γιατί αυτό μπορεί να γίνει μόνο σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Άρα οι δυνάμεις ασφαλείας ε, είναι ένα σημαντικό τμήμα των υπηρεσιών που υποτίθεται ότι πρέπει να παρέχει το κράτος. Όσον αφορά τώρα την Αφρικανική Ένωση, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η Αφρικανική Ένωση είναι μια βραχυπρόθεσμη λύση. Όταν αποφασίστηκε από την, από την Αφρικανική Ένωση ότι θα παρέμβουν πριν από μερικά χρόνια, ήταν μία από τις αρχές, οι αρχές, μία από τις αρχές του ήταν, θα ήταν βραχυπρόθεσμη επέμβαση, όχι μακροπρόθεσμα. Ε, όπως ήταν η περίπτωση του Σουδάν για παράδειγμα, κατά κάποια στιγμή, κατά κάποια στιγμή θα αντικατασταθούν οι δυνάμεις από τον ΟΗΕ. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ο ΙΕ θα κάνει οτιδήποτε στη Σομαλία μετά από την τελευταία του προσπάθεια στην περιοχή. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μια, εθνική, ε, μια ανάπτυξη εθνικής ασφάλειας στη Σομαλία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Μπραντνερ. Έχω δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις μιλάτε για εκπαίδευση 3.000 ατόμων, μιλήσετε για 800 στρατιώτες. Πόσοι είναι στρατιώτες, πόσοι είναι αστυνομία, πόσοι είναι συνοριοφυλακοί. Ποιος που θα εκπαιδευτεί, ποια κατηγορία εκπαιδευτικού προσωπικού χρειάζεται. Δεύτερον, γιατί να μην αφήσουμε τους Γάλλους να συνεχίσουν και θέλουν οι Γάλλοι να συνεχίσουν. Δεν ξέρω αν υπάρχει κανένας Γάλλος στην αίθουσα για να απαντήσει, αλλά εν πάση περιπτώσει... Ενδεχομένω να έπρεπε να αφήσω πρώτα του Γάλλου να απαντήσουν και μετά να πάρω εγώ το λόγο, λέει ο στρατηγό Ζωανά. Εντάξει. Αν δεν υπάρχει κανεί εγώ θα διαβιβάσω τις ε, ερωτήσεις σας. Κοιτάξτε, για το στόχο 5.000 ε, στρατιωτικές δυνάμεις ε, είχαν απαντήσει οι ίδιοι Σομαλοί ότι χρειάζονται. Αυτή τη στιγμή όμως ε, η δουλειά που κάνει το εργαστήριο αξιολόγησης δεν έχει καταλήξει ακόμη πουθενά, δεν έχουμε τα συμπεράσματα της εργασίας αυτής. Σε πρώτη φάση νομίζω 6-7 άτομα θα είναι και 10.000 αστυνομικοί ε, που θεωρούνται απαραίτητοι για την, ασφάλεια, την εξασφάλιση ε, της ε, ασφάλειας της μεταβατικής κυβέρνησης. Στη, στο Μογκαντήσου αυτή τη στιγμή νομίζω 752, 752 έχει μετρήσει η κυβέρνηση στο Μογκαντήσου. Δεν ξέρω βέβαια τώρα, ίσως είναι λίγο πρόχειρα τα ε, αριθμητικά μου στοιχεία. Μου φαίνεται 500-600 εκπαίδευσαν οι Γάλλοι, 862 η Ουγγάντα, 2.000 με 2.500 παραμένουν ανεκπαίδευτοι. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να, μπορούν να συμμετέχουν και άλλοι στην εκπαίδευση. Είναι μια αποστολή που ουσιαστικά δεν σημαίνει πάρα πολλά πράγματα και υπάρχουν ακόμη τάγματα ε, περίπου 2-3 χιλιάδων που πρέπει ακόμη να 2-3 τάγματα που, που πρέπει ακόμη να εκπαιδεύσουμε. Επίσης πρέπει να δούμε και τα θέματα του εξοπλισμού, των μισθών, ε, του ανεφοδιασμού των ε, στρατιωτών όταν βρίσκονται στη Σομαλία. 2.000 άτομα περίπου, όπως είπα και προηγουμένως. Αλλά είναι χοντρικός υπολογισμός. Ε, θα είμαστε πιο ακριβείς στη συνέχεια. Να απαντήσω και για την Ερυθρέα. Κοίταξε, εγώ δεν είμαι ιδιαίτερα ειδικό για το θέμα τη Ερυθρέα. Όσον αφορά τώρα την αλλαγή, την πολιτική, κανεί δεν μπορεί να το πει αυτό ότι θα γίνει με βεβαιότητα. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο μας υποδέχτηκαν, ε, ο τόνος της συνομιλία με τις αρχές της Ερυθρέα, δείχνει ότι καταρχά είχαν ανάγκη να μιλήσουν, να τα βγάλουν από μέσα του ενδεχομένως να είναι και προσωπική μου ερμηνεία, είναι υπό την απειλή των ε, κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ε, και είναι κάπως υποχρεωμένοι να πούν αυτά που θέλουν ε, να πούν από εκεί και πέρα τους ε, ενδιέφερε πάρα πολύ το μέλλον του Σουδάν γιατί είναι ένας αποσταθεροποιητικός παράγοντας και για το μέλλον της Σομαλίας. Οπότε έχω την εντύπωση ότι για αυτή την ε, χώρα που μοιάζει με τη Βόρεια Κορέα, δεν έχω πάει ποτέ, ε, με την Αλβανία ίσως μοιάζει επίσης, αλλά εκεί έχω πάει, ενδεχομένως 10 χρόνια απομόνωσης πέρασαν και θέλουν κάποια διέξοδο. Δυστυχώς όμως έκλεισαν όλες αυτές τις πόρτες γιατί κατά κάποιο τρόπο τους έχουν ε, εγκαταλείψει στη μοίρα τους. Οπότε θέλουν πάρα πολύ να συμμετέχουν σε ένα διάλογο. Τώρα από εκεί και πέρα κατά πόσο θα χειραγωγηθεί αυτός ο διάλογος ε, ή αν πρόκειται να συνεχιστεί ή τέλος πάντων είναι απολύτως ειλικρινής δεν το ξέρω, θα το δούμε στο μέλλον αλλά είναι γεγονός ότι δεν πρέπει να κλείσουμε την πόρτα και νομίζω το είχε πει και ο πρέσβης εδώ πριν από τρεις εβδομάδες ότι Πρόκειται για μια μεταβατική κυβέρνηση την οποία δημιούργησε η διεθνή κοινότητα και την οποία υποστήριξε η Αφρικανική Ένωση προσπαθώντας ε, να ε, καταπολεμήσει ουσιαστικά τον ίδιο τον πληθυσμό της Σομαλίας. Όχι, εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, προφανώς. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά το ερώτημα της ε, υποφορά την θέληση των Γάλλων, μπορούμε αύριο το βράδυ να θέσουμε το θέμα στον Σουηδό Υπουργό Αμήνης, ε, στη σύνθεση των Υπουργών Εξωτερικών, ε, ο οποίος άλλωστε θα προεδρεύσει τη συνεδρίαση αυτής ενδεχομένως να μπορεί να σας πει ορισμένα πράγματα. Δεν είμαι και πάρα πολύ σίγουρος ότι υπάρχει τέτοιου είδους ε, θέληση παρέμβασης ε, των, ε, από πλευράς Γάλλων. Αυτό που γνωρίζουν ότι υπάρχει μια θέληση προβληματισμού για το πώς θα είναι μια αμοιβαία προσπάθεια και υποστηρίζοντας βέβαια τη διαδικασία του Τζιμπούτι, Το είπατε και εσείς ότι ο πολιτικός στόχος είναι να υποστηρίξουμε την Αφρικανική Ένωση σε μια διαδικασία η οποία έχει διεθνώς αναγνωριστεί και η οποία καρποφορεί θα λέγαμε από απόψε ως πολιτική σταθερότητα. Έχουμε μια μεταβατική κυβέρνηση η οποία εντάξει δεν είναι τέλεια αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αντικείμενο κάποια συνένεση εν πάση περιπτώσει που δεν ίσχυε για τις προηγούμενες προσπάθειες, με τις προηγούμενες προσπάθειες που είχαν γίνει. Ε, τώρα όσον αφορά πολιτικές προτεραιότητες μπορούμε να, να, να, αναρωτηθούμε όσον αφορά και τις γεωπολιτικές αλλά και τις γεωγραφικές μας ε, ε, προτεραιότητες. Ένας από τους βασικούς μας στόχους ε, είναι να αποφύγουμε η Σομαλία που είναι ήδη σε μια κατάσταση όχι πάρα πολύ καλή, να μην γίνει ένα μελλοντικό Αφγανιστάν και η εσωτερική αστάθεια που εξακολουθεί να υπάρχει σε ορισμένες περιοχές να μην εξαχθεί όπως γίνεται ήδη μέσω του φαινομένου που δεν αναφέραμε των προσφύγων γιατί υπάρχει ροή προσφύγων ε, προς το Τζιμπούτι, προς την Κένια ε, πήγαμε κιόλα και είδαμε ότι είναι πολύ ανησυχητικά τα πράγματα όσον αφορά λοιπόν τη σταθεροποίηση της κατάστασης Εντάξει, υπάρχουν πολλά ερωτήματα και μπορούμε να αναρωτηθούμε για την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης και των αστυνομικών και των στρατιωτών ε, ε, προς όφερος Ομαλίας. Αυτό είναι το πλαίσιο λοιπόν του προβληματισμού μας. Ο κύριος Μπούτι Κόφερ και μετά θα ολοκληρώσουμε να συγκρίνεται και πάλι τη Σομαλία με το Αφγανιστάν και ίσως αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πιο ενδελεχώς. Εγώ όμως αναρωτιέμαι αν με τέτοιου είδους δέσμευση έναντι της προσωρινής κυβέρνησης στη Σομαλία μήπως ποντάρουμε σε μια εξουσία η οποία είναι φανερό ότι είναι ακόμα λιγότερο σε θέση να δώσει προοπτικές σε αυτή τη χώρα από ό,τι μπορούμε να πούμε για την αντίστοιχη κυβέρνηση στο Αφγανιστάν. Η δημιουργία κράτους στο Αφγανιστάν είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα. Παρ' όλα αυτά, το 1 τρίτο περίπου των Αφγανών, όπως φαίνεται από τις εκλογές, παρά τις απάτες και τις ατασταλίες, υποστηρίζει αυτό το εγχείρημα. Εγώ φαντάζομαι Σομαλία ούτε καν μπορεί να φανταστεί κανείς να έχει μια εκλογή που να έχει συμμετοχή του ενός τρίτου του πληθυσμού. Τι είναι αυτό το οποίο μας νομιμοποιεί αυτή την ενέργεια μια κυβέρνηση μεταβατική, η οποία με χίλιου στρατιώτε να την υποστηρίζει ότι όλα αυτά θα συμβάλλουν σε μια πραγματική προσπάθεια δημιουργία κράτου. Πολύ ωραία είναι στα χαρτιά των να φτιάχνουμε κράτη, αλλά στην πράξη να έχουμε ένα κράτο το οποίο αυτή τη στιγμή βασίζεται σε μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει καμία ρανίδα εξουσία έξω από το Μογαδίσιο, αυτό είναι μια χήμερα τελείω. είναι μια τρέλα. Ο κύριο Γιάννη. Δεν ήθελα να παρέμβω σε αυτή τη συζήτηση. Το είχε κάνει νομίζω υποφελώ ο συντονιστή τη ομάδα μα, ο Ρομπέρτο Γκουαλτιέρη. Εγώ μετά από όλες αυτές τις ερωτήσεις, εγώ συμμερίζομαι απόλυτα τον σκεπτικισμό που έχουν αναφέρει όλοι οι συνάδελφοι. Οι δυνατότητες επιτυχίας ναι μεν είναι πάρα πολύ περιορισμένες, αλλά εγώ δεν βλέπω άλλη εναλλακτική λύση από την αδράνεια και αργία μη την κακίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά την διάσταση άμυνας και ασφάλειας δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζει καταστάσεις τόσο μεγάλης δυσκολίες. Αλλά το να κάνουμε μια προσπάθεια να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια και την σταθερότητα που εναπόκειται καταρχήν στους Σομαλούς φυσικά και να αποφύγουμε τις πειρατικές δράσεις. Όλα αυτά είναι κάτι το οποίο εγώ πιστεύω ότι είναι ένα αξιόλογο εγχείρημα και αξίζει την υποστήριξή μας. Θα δούμε στο μέλλον πώς θα εξελιχθούν αυτά τα πράγματα, αλλά θέλω και εγώ να υποστηρίξω και τον Πρόεδρο σε αυτά που είπε. Ευχαριστώ. Μήπως η Κομισιόν θέλει να πάρει το λόγο. Δύο λογάκια μόνο. Γιατί είναι θεμητό το ερώτημα. Τι νομοποιεί αυτή τη μεταβατική κυβέρνηση. Δύο πραγματάκια λοιπόν σημαντικά. Πρώτα απ' όλα αντιλαμβάνεστε πως ε, είναι μία σύγκρουση μεταξύ φυλών. Πρόκειται περί τεσσάρων φυλών που βρίσκονται σε πόλεμο 17-18 χρόνια. Και οι Κομισιόν και άλλοι προσπάθησαν να βρουν τρόπους να σταματήσει η σύγκρουση και να υπάρξει κάποια τάξη. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει κάποιο είδου κυβέρνηση. Οπότε δεν είναι τώρα ώρα για εκλογές. Και γεννήθηκε από μια διάσκεψη η κυβέρνηση. Μια διάσκεψη που χρηματοδότησε και υποστήριξε η Κομισιόν. Κράτησε ένα χρόνο, ίσως και παραπάνω. Και η διάσκεψη έφερε εκπροσώπους όλων αυτών των φυλών από κάθε, κάθε φατρία και υπάρχει λοιπόν μία εκπροσώπηση όλων αυτών στην μεταβατική κυβέρνηση για να αποκατασταθεί κάποιο είδους νόμος και τάξη για να οδηγηθούμε σε εκλογές. Αυτή είναι η νομοποίηση αυτής της κυβέρνησης. Προέκυψε μέσω των διαπραγματεύσεων, μέσω των φαντριών αυτών και προσπαθήσαμε να φέρουμε και αντιφρονούντες για να γίνει πιο, αποτελεσμα... πιο αντιπροσωπευτική όσο περνά ο χρόνος. Θεμητό αυτό που λέτε λοιπόν, αλλά υπάρχει κάποιος βαθμός νομοποίησης. Και ούτω ή άλλω υποτίθεται ότι είναι μεταβατική κυβέρνηση. Ευχαριστώ. Θα συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να θέσουμε και ερωτήματα αν θέλουμε στον Υπουργό Άμυνα της Σουηδίας από τις 6.30. Σε ό,τι αφορά την υποεπιτροπή μας, η επόμενη